Dear colleagues, I'm going to make a prompt start today because we have less than an hour for the president. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε αμέσω ε, γιατί ε, έχουμε λιγότερο από μία ώρα για το θέμα που αφορά στην Προεδρία. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε πάρα πολύ, διότι είμαι σίγουρος ότι θα υποβληθούν πολλές και καλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήρθατε στην ώρα σας, όσοι ήρθατε στην ώρα σας και θα ήθελα να ξεκινήσω με την έγκριση της μερίσια διάταξης και να προτείνω τις εξής αλλαγές. Το 3 πάει για το Σεπτέμβρη. Το 15 θα λάβει χώρα ε, στις 12 ε, Ιουλίου, το 16 θα μοιραστεί ανάμεσα στις προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας τον κύριο Αντρές Άμπελ που είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε και αυτό θα γίνει τώρα. Τώρα δηλαδή. μέσα μετά αυτέ τις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Και το 16 ε, επίσης ε, ε, θα αφορά στις, προ... στις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας ε, σχετικά με την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 17 αναβάλλεται το Σεπτέμβρη και θα έχουμε ένα νέο σημείο 17 σχετικά με το θέμα των καταγγελόντων. Εάν λοιπόν δεν έχετε αντιρρήσεις ε, θα έλεγα να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Και τέλος, ε, επιτρέψτε μου να κάνω και κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Δεν θα έχουμε μαλτέζικα, κροατικά και γκέλικ. Και επίσης ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ θα είναι ο εισηγητής για τους ε, τον έλεγχο των ε, ρευστών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνείτε από ό,τι βλέπω, ναι. Οι ε, εφαρμοστικέ και εκτελεστικέ πράξεις είναι το σημείο 3 των ανακοινώσεών μου και κατόπιν όσον αφορά την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Αυτό αφορά ε, τις πρόδρομες ουσίες. Στις 11 ε, Απριλίου συζητήθηκε αυτή η έκθεση και της Επιτροπής και το άρθρο 14.2 του κανονισμού απαιτεί ε, να ε, γίνει εκχώρηση αρμοδιοτήτων για πέντε χρόνια από τις 1η Μαρτίου και θα υπάρχουν άλλα εννέα μήνες ε, πριν από, το τέλος περίοδου. Μιλάμε για μια ταυτόσιμη διάρκεια, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αντιδράσει στην παράταση πριν από το τέλος περίοδου. Στην περίπτωση που ε, το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει με αυτή τη σιωπηρή παράταση, σιωπηρή λοιπόν παράταση, ε, τότε θα πρέπει να εγκρίνει ένα ψήφισμα που θα είναι κατά της παράτασης και αυτό μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2017. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω μια καταληκτική ημερομηνία έτσι ώστε να μπορεί να κατατεθεί αντίδραση από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής μέχρι τις 11 ε, Σεπτεμβρίου του 2017, τις 12 ώρα το μεσημέρι. Ε, από ό,τι βλέπω δεν πολύ παρακολουθείτε. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία αύριο στις 5.30 και την Τετάρτη στι 10 και 4 το πρωί. Ε, αν έχετε καλοσύνη να έχετε μαζί σα ε, τις κάρτες σας για να μπορείτε να ψηφίσετε. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο, το νέο τρία και είναι η παρουσίαση από τον κύριο Άντρε Ανβελτ, ο οποίος είναι υπουργό Ετορικών της Δημοκρατίας της Εστονίας. Σας καλωσορίζουμε θερμά κύριε Ανβελτ και χαιρόμαστε που σας έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της εσθονική Προεδρίας. Αυτή είναι η πρώτη σας ε, εισήγηση στην Επιτροπή μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν ιδιαίτερα θερμά. Και πριν ε, αναφερθώ στην πρακτική οργάνωση της σημερινής συνεδρίασης, θα ήθελα να αναφέρω ότι ε, το άτυπο συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας στο Ταλίν. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και ευχαριστώ πολύ εσάς ε, και την ομάδα σας για την προετοιμασία. Απλά να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι ε, θα ακούσατε σχετικά με τα στρατηγικά σημεία της Εστονικής Προεδρίας, τι θέλει να κάνει η Εστονική Προεδρία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται στην ε, συνάντηση όσον αφορά τα θέματα της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων. Τα στοιχεία κλειδί, αυτά που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, είναι η ε, η τοποθέτηση σχετικά με τη Λιβύη και τη Μεσόγειο. Αυτό είναι ένα θέμα που κυριαρχεί και ξέρω ότι ο Υπουργό Εσωτερικών θα θελήσει να μιλήσει για αυτά τα δύο κομβικά θέματα, όπως και για ευρύτερα στρατηγικής φύσεως θέματα. Δεν θέλω να καταναλώσω άλλο από τον χρόνο σας, ε, θα ήθελα όμω να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή αρχή στην Προεδρία με αυτή την άτυπη συνάντηση. Και αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο για αυτήν, θα ακούσετε και άλλα στοιχεία τώρα που θα ε, μιλάει. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τον κύριο Άνβελτ να μιλήσει για 10-15 λεπτά και μετά οι συνάδελφοι θα υποβάλουν ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλώ ενώπιον σας σήμερα η Εσθονία Ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από δέκα μέρες. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για την πρώτη Προεδρία την οποία, ε, ε για την οποία επιφορτίζεται η χώρα μου τόσο ο λαός όσο και οι αρχές και η κυβέρνηση κατανοούν την σημασία αυτής της ε, ευθύνης. Οπότε αφενός ε, ε, χαιρόμαστε που αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση, ε, αφετέρου θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Όταν η Εστονία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004. Θυμάμαι στην Εστονία ήταν μια πολύ όμορφη ανεξιατική μερα και ο λαός ήταν γεμάτος από χαρά, γαλίαση και αισιοδοξία. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είχαν διαρκέσει 6,5 χρόνια. Τέσσερα χρόνια μετά γίναμε πλήρη μέλη της ζώνης Σέγγεν, ε, δεν γίνονται έλεγχοι στα σύνορά μας, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και στα χερσαία σύνορα πλέον. Όλοι μας λοιπόν αναγνωρίζουμε τη σημασία της ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρώπη. Ε, πέρασαν 9 χρόνια και κάτι μήνες από τότε, ε, γεμάτα ε, τραχώδη χρόνια για όλους μας. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρώπη επλήγει από, την κρίση ευρωζώνης, ε, την οικονομική ε, και τραπεζική κρίση, την μεταναστευτική κρίση, ε, τα προβλήματα στην γεωργία. Ε, η καθημερινότητα πλέον δεν είναι όπως ε, διαμορφωνόταν όταν εμείς μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στην Εστονία είμαστε ακόμα πιο προσιλωμένοι στο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις, να φέρουμε σε πέρα τις ευθύνες μας με έναν τρόπο συνετό. Αυτό άλλωστε πρέπει να κάνουν και όλες οι προεδρίες. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις. Εγώ είμαι υπεύθυνο για την μετανάστευση, το άσυλο ε, και, τις, ε, για τους συνορικούς ελέγχους, καθώς επίσης και για την εσωτερική ασφάλεια, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα θέματα προκύψουν επίκαιρα. Κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου και την εφαρμογή του, της εντολής για την υπηρεσία ελέγχου των ε, συνόρων χερσαίων και θαλασσίων συνόρων. Ε, θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα στο μυαλό μας τα προβλήματα στη Μεσόγειο και πιο πολύ στην κεντρική Μεσόγειο. οι Ιταλοί συνάδελφοι θα χρειαστούν τη στήριξή μας οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων στο Τάλιν τον ε, Ιούλιο ε, συζήτησαν πώς μπορούν να στηρίξουμε την Ιταλία περισσότερο. Ε, το Κορεπέρ στις 12 Ιουλίου μάλιστα θα συζητήσει ξανά αυτό το θέμα. Η ασφάλεια των πολιτών μας είναι εξίσου σημαντική. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την αίσθηση της ασφάλειας. Τα συστήματα πληροφόρησης και η διαλειτουργικότητά τους είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, και αυτό το λέμε εδώ και χρόνια. Στην Εστονία ε, η διαλειτουργικότητα έχει επιτευχθεί εδώ και πολύ καιρό ήδη. Και μάλιστα υπερβαίνει τον τομέα των, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων και η διαλειτουργικότητα του σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί θα βελτιώσει την δυνατότητα των κρατών μελών να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και την γενικότερη ασφάλεια στις χώρες μας. Διαλειτουργικότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να απαλληφθούν τα τεχνικά εμπόδια ε, που, ε, στην πρόσβαση αυτών που έχουν το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να ε, συμβολεύονται αυτά τα στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ούτε ότι θα πληγούν τα προσωπικά δικαιώματα. Ε, αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπάρχουν πολλές διαπραγματευτικές προτάσεις και είναι πολύ σημαντικό κανείς να έχει ε, προτεραιότητες, ε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια χώρα μικρή όπως η Εστονία. Όμως, ε, <laughs> η πραγματικότητα είναι ότι όλα είναι προτεραιότητες. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Πριν περάσω στις συγκεκριμένες προτάσεις, θα ήθελα να πω ότι ο Εστονός Υπουργός ε, Δικαιοσύνης ε, θα βρεθεί εδώ μπροστά σας αύριο για να σας ενημερώσει για τις δικές του ευθύνες. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Κυρίε και κύριοι. Τα θέματα σχετικά με την μετανάστευση βρίσκονται στην, ε, στο, στην πρώτη θέση της ημερήσιας διάταξη εδώ και τα πολλά κάποια χρόνια. Η Στονική Προεδρία θα συνεχίσει την δουλειά που έχει ήδη ξεκινήσει και είναι επίγουσα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα της μετανάστευσης. Ε, η, Προκλήσεις είναι πολλέ, αλλά ο στόχο μα είναι σαφή. Θέλουμε σταδιακά να θέσουμε σε εφαρμογή ένα κατάλληλο και δίκαιο ε, σύστημα ασύλου και μεταναστευτική πολιτική ο ακρογωνίος λίθος αυτών των πολιτικών θα πρέπει να είναι ο αποτελεσματικό έλεγχος των εξωτερικών μας συνόρων. Μακροπρόθεσμα μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μέσο πρόθεσμα και βράχη πρόθεσμα μέτρα τα οποία ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Θα συνεχίσουμε την εργασία που έχει ήδη ξεκινήσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι για να πετύχουμε θα πρέπει ε, να ε, προχωρήσουμε παράλληλα όλα τα ζητήματα και ε, όλες τις συνιστώσεις. Η Ελλάδα και η Ιταλία ε, ιδιαίτερα ε, βρίσκονται στο μέτωπο του αγώνα αυτού. Χιλιάδες παράτυποι μετανάστες φτάνουν κάθε μήνα. Αυτό απαιτεί να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση καθώς επίσης και την παροχή ε, εμπειρογνωμόνων ε, από την Υπηρεσία Ασύλου και τη Frontex. Η Προεδρία καλωσορίζει το πρόγραμμα δράσης Κομισιόν για να στηρίξει την Ιταλία που υιοθετήθηκε στις 4 Ιουλίου και συζητήθηκε στο Τάλιν κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 6 και 7 Ιουλίου. Ε, θα ακολουθήσουμε, θα πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να ξεκινήσει να εφαρμόζεται γρήγορα το σχέδιο. Αυτή την εβδομάδα μάλιστα θα συζητηθεί σε διάφορα φόρουμ. Σκύφα, Κορεπέρ, στην IPCR, στο, στο, Στρογγυλή Τράπεζα Υψηλού Επιπέδου κλπ. Τον περασμένο Φλεβάρι στη Μάλτα οι ηγέτε μα συμφωνήσαν πώ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κατάσταση στην κεντρική Μεσόγειο και να μειώσουμε ε, τον αριθμό των παράνομων διαβάσεων παράτυπων διαβάσεων, συγγνώμη, ε, να διακόψουμε, να διαρρήξουμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο ε, των συμμοριών ε, και των λαθρεμπόρων και να σώσουμε ζωές στη θάλασσα. Ε, βασιζόμενοι στη, στην δήλωση της Μάλτας, η Μαλτέζικη Προεδρία ετοίμασε ένα σχέδιο δράσης και εμείς θα το συνεχίσουμε. Η αποτελεσματική πολιτική επιστροφών ε, είναι σημαντικό τμήμα της πολιτικής μετά σε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη επιτυχία να μειώσουμε, για προκειμένου να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου ε, σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Η δική μας προθέση είναι να επενδύσουμε περισσότερο στο να ε, βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής επιστροφών αντιμετωπίζοντας και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πτυχές της. Χρησιμοποιώντα το σύστημα ε, πληροφοριών Schengen για, την, ε, για διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι αποφάσει επιστροφή, μπορεί να θεωρηθεί ένα σημαντικό βήμα προ αυτήν την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση ε, έχουμε δει σημαντική πρόοδο τελευταία. Ε, πάνω από 20.000 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι με πρόσθετες προσπάθειες ε, είναι ακόμα δυνατό να μετεγκαταστήσουμε και τους υπόλοιπους υποψηφίους προς κατάσταση που βρίσκονται στην Ιταλία και την Ελλάδα. Εξακολουθούμε να ε, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, θα φέρουν σε πέρας τις ευθύνε τους και ότι θα μετεγκαταστήσουν τις, τους, τις ποσοστώσεις τους έγκαιρα. Σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση βρισκόμαστε στα δύο τρίτα του στόχου που είχε τεθεί μεταξύ των 21 κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νόμιμη ε, μετανάστευση, ε, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε ε, την δυνατότητά μας να προσελκύσουμε υπηκός τρίτων χωρών με τα κατάλληλα προσόντα. Η διοδηγία μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια της προτεραιότητας της Προεδρίας μας λοιπόν. Θέλουμε να ξεκινήσουμε ε, διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για αυτό το θέμα. Αλλά να υπογραμμίσω ότι σύμφωνα με τις ε, απόψεις που ακούγονται στο Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να εκδίδουν άδειε μόνιμης κατοικίας, και μόνιμης κατοικίας για τους εργαζόμενους που έχουν ψηλά προσόντα και σύμφωνα με τον εθνικό τους δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την πολιτική θεωρήσεων, ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον κώδικα θεωρήσεων. Ε, θα πρέπει η συζήτηση να αποσυνδεθεί από την, το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων μετά θα περάσουμε σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Αν συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση, ε, θα ζητήσω από την ομάδα μου να ξεκινήσουν τεχνικέ εργασίε ε, μαζί με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε, για να δώσουμε, για μάλλον να καθισκάσουμε το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Η Εστονική Προεδρία ε, εργαζόμενοι πάνω στην ε, δουλειά που ε, έφεραν σε πέρα στι προηγούμενε προεδρίε κάτω χώρε Σλοβακία και Μάλτα θα συνεχίσει την εξέταση όλων των νομοθετικών προτάσεων σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματο ασύλου. Θα κάνουμε ό,τι πάνε από το χέρι μα για να πετύχουμε όσο δυνατό περισσότερη πρόοδο σε ό,τι αφορά τα διάφορα ζητήματα του συνολικού πακέτου μεταρρύθμιση. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη τη ε, υπηρεσία εξωτερική δράση σε μια συγγνώμη, του οργανισμού ασύλου σε μια ε, υπηρεσία ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα με το Κοινοβούλιο από το Γενάρη. Ε, έχει, έχουν γίνει διάφορες συνδέσεις του τριμερούς διαλόγου, τεχνικές συναντήσεις κλπ. και έχει γίνει γενικά σημαντική πρόοδος. Παρ' όλα αυτά ε, θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά κατά τη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά τη Eurodac, το Συμβούλιο ε, κατέληξε μια μερική γενική ε, προσέγγιση το περασμένο Δεκέμβρη. Η Προεδρία τη ε, Μάλτα διεύρυνε την εντολή του Συμβουλίου ακόμα περισσότερο, αλλά ορισμένα θέματα εξαρτώνται από άλλε σχετικέ προτάσει που εκκρεμούν. Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του Δουβλίνου θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να βρούμε ένα συμβιβασμό για το πώς θα εφαρμοστούν οι αρχές της ευθύνης και της αλληλεγγύης. Κατά διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι υπουργοί και πρέσβεις ε, ε, συζήτησαν το θέμα αυτό. Ορισμέ... Κάποιος κοινός παρανομαστής σε ό,τι αφορά ε, ορισμένες πτυχές ε, αλλά χρειάζεται περισσότερη πρόοδο σε άλλα σημαντικά θέματα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έχουν λάβει η χώρα, υπήρξε ευρεία στήριξη για μια ε, ολιστική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος κανονισμός ε, του Δουβλίνου και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου είναι κομμάτια ενό ε, μεγαλύτερου πάζλ. Οπότε και η μεταρρύθμιση θα πρέπει να επιδιωχθεί παραλλήλου με άλλες πολιτικές, μεταξύ άλλων ε, η καταπολέμηση των ροών παράτυπης μετανάστευσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ενίσχυση των επιστροφών ε, και να δούμε πώ θα διασφαλίσουμε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι στα σύνορα θα παραμείνουν η εξαίρεση. Η Ιστονική Προεδρία δίνει μεγάλη σημασία στην εξέταση όλων των προτάσεων του δεύτερου νομοθετικού πακέτου τη μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου. Σημαντική πρόοδο έχει σημειωθεί σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά την πρόταση ε, κανονισμού για τις προποθέσεις της χορήγησης ασύλου. Βάσει των εργασιών τη Μαλτέζικη Προεδρία και εμεί ελπίζουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτή την πρόταση και να ξεκινήσουμε τι συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα επιδιώξουμε την εξέταση ε, τη οδηγία περί προποθέσεων υποδοχή ε, και του ευρωπαϊκού πλαισίου ε, επανεγκατάσταση ε, και αν αυτό καταστεί δυνατό θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξαιτία τη πολυπλοκότητα του φακέλου δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο ό,τι αφορά τον κανονισμό περί διαδικασία ασύλου και ελπίζουμε να συνεχίσουμε την εξέταση σε τεχνικό επίπεδο. Όπω γνωρίζετε, οι συνομοθέτε έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τι διαπραγματεύσει για την πρόταση κανονισμού για τι ασφαλεί χώρε προέλευση και εξακολουθούν να επεξεργάζονται αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του κανονισμού διαδικασίας ασύλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια, δυστυχώς ε, είδαμε και τις πρόσφατες ε, πολύ άρθμες τρομοκρατικές επιθέσεις και έτσι καταλαβαίνουμε ότι συγκολουθεί να υπάρχει η απειλή του, της τρομοκρατίας. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν τον περασμένο μήνα καλούν για ανάληψη συγκεκριμένη δράση ό,τι αφορά την ε, κατά της τρομοκρατίας, του μίσους και του βίαιου εξτρεμισμού. Επομένω, θα κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μα για να περιορίσουμε και να καταπολεμήσουμε αυτή την απειλή. Ε, Όμω, απαιτείται ένα μακρόπνο σχέδιο, προσήλωση και ε, συνεχεί προσπάθειε με Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, αλλά και από τον κλάδο και του παρόχου ε, υπηρεσιών για την καταπολέμηση ε, τη ε, επιγραμμική τρομοκρατία. Στο ε, Συμβούλιο Αστυνομικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνη του Ιουνίου, οι Υπουργοί χαιρέτησαν τη θέσπιση ε, μιας ε, ομάδας ψηλού επίπεδου για την ριζοσπαστικοποίηση. Ως Ένωση έχουμε σαφή ε, νομική και ηθική υποχρέωση να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Ξέρετε τις συνεχόμενες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα όπως είναι οι αλλοδαποί μαχητές και το καθεξής. Εργαζόμαστε σκληρά λοιπόν για να ελοποιήσουμε αυτά τα μέτρα και παρότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πάντα υπάρχει σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά και τι ενωσιακέ βάσει δεδομένων. Ε, είμαστε απόλυτα προσελωμένοι στη συνέχιση και στην προώθηση του συστήματος ε, ε, πληροφοριών Schengen που παρουσιάστηκαν το 2016 από την Επιτροπή. Αυτές οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν αλλαγές που θα μας βοηθήσουν κατά πολέμου στην δημοκρατία, εισάγοντα και μια υποχρέωση δημιουργία μιας ενό alert, μιας επισήμανσης ε, εσεί, σε περιπτώσει που συνδέονται με τρομοκρατικά δικήματα, ε, σε μια νέα διαδικασία που θα επιτρέψει στι αρχές να συλλέγουν πληροφορίε. Η Προεδρία θα συνεχίσει να εξετάζει αυτές τις προτάσεις ε, κατά προτεραιότητα. Βάσει των συζητήσεων που έλαβαν υπόψη ε, τον Ιούνιο, ε, ο σκοπός μας είναι να πετύχουμε γενική προσέγγιση το φθινόπωρο. Μετά θα είμαστε σε θέση επιτέλους να ξεκινήσουμε τουλάχιστον τις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις στα τέλη του 2017. Προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, έχει σημειωθεί ένα σημαντικό πρωτοβήμα με τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης του συνοριακού κώδικα Σέγγεν, που παρέχει και προβλέπει μάλλον συστηματικούς ελέγχους στα εξωτερικά μα σύνορα. Η πρόσφατη συμφωνία στα πολιτικά ζητήματα στο σύστημα εισόδου-εξόδου ήταν ακρογωνία λήθο για την επίτευξη μια συμφωνία, ε, ελπίζουμε ήδη αυτή την Τετάρτη. Η επίτευξη μια πολιτική συμφωνία σε άλλου φακέλου, ε, όπω το σύστημα αίτια και στο σύστημα ΣΥΣ, ε, θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. προτεραιότητα για μας είναι και το Ευρωπαϊκό ε, Σύστημα Πληροφοριών ε, Αίτιας. Τώρα που καταφέραμε να ε, καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση, θα ξεκινήσουμε τη πραγματεύσει με το Κοινοβούλιο των Σύμμετρο Δυνατών, προκειμένου να πετύχουμε συμφωνία μέχρι τα τέλη της Προεδρίας μας. Η Προεδρία επίση θέλει να εργαστεί για την διασφάλιση τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων για την διαχείριση συνόρων, τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Το Συμβούλιο χαιρέτησε τις συστάσεις από την ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας. Από το φθινόπωρο και μετά η Προεδρία είναι διατεθειμένη να εργαστεί μαζί σας αλλά και με την Επιτροπή για να προετοιμάσει το έδαφος για τις ε, επερχόμενες προτάσεις ε, διαλειτουργικότητας. Σκοπός μας είναι να άρουμε τεχνικά εμπόδια από τα δεδομένα που ήδη συλλέγουμε και να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρον. Και έτσι, αν κάνουμε καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεδομένων, δεν θα χρειαζόμαστε να συλλέγουμε όλα και περισσότερα δεδομένα. Βέβαια, αυτό δεν θα έχει καμία ε, ε, επιρροή στις συνεχόμενες εργασίες για τις νομοθετικές προτάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στο αίτια, στο ΣΥΣ και το καθεξής. Για τη λειτουργικότητα πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των ε, ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι θέματα βασικής προτεραιότητας. Και για μας τους εστονούς είναι πολύ σημαντική διαλειτουργικότητα και η πληροφορική, ακριβώς επειδή παρέχει και δεδομένα, προστασία δεδομένων υψηλού επίπεδου, αλλά και διαφάνεια στην χρήση των δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατάλληλη εντολή για να υλοποιήσουμε ε, τις ε, πρακτικές αυτές ε, διαλειτουργικότητας στην πράξη. Επίση, θεωρούμε ότι και η πρόταση για την EU Λύσα είναι θέμα προτεραιότητα για την Προεδρία μα, προκειμένου να πετύχουμε γενική ε, προσέγγιση μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Κυρίε και κύριοι αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ ε, και μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω τι προτεραιότητε τη Εστονικής ε, Προεδρία προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί ένα ασφαλή χώρο για του ε, πολίτε μα και του επισκέπτε μα Είμαι στη διάθεσή σα για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριο Μωράς. Δεν ξέρω τι συνέβη με τα φώτα. Ελπίζω να μην φταίνουν οι Ρώσοι. Μήπως μακρηγόρησα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέει ο Πρόεδρος. Το πρόβλημα είναι ότι το θέμα είναι ότι έχουμε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που περιλαμβάνει τόσους πολλούς ε, φακέλους και έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας ε, για έναν μεγάλο αριθμό και ένα ευρύ φάσμα περίπλοκων ζητημάτων. Η συνάδελφος στήσει το λόγο. Τέσσερις προς το παρόν μόνο. Σίπελ, Γκόμες, Γιόρκ και Κοέλιο. Μπορείτε να μου πείτε, παρακαλώ πείτε μου αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Για όσους έφτασαν μόλις, αναφέραμε εισαγωγικά ότι το άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνη Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το θέμα της Λιβύης, αλλά υπήρχαν και άλλα στρατηγικά ζητήματα που ανέφερε και ο Υπουργό ε, και μπήκαν στην μέσα όπως το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας, το αίτιας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καλύψουμε όλα σήμερα. Ήθελα μόνο να αναφέρω το θέμα που αποτελεί προτεραιότητα, αυτό της Λιβύης και το σχέδιο εργασίας ε, της Επιτροπής καθώς και ο κώδικας δεντολογίας. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί με ζητήματα ασύλου και άλλα θέματα. Το ανέφερα και στον ε, Υπουργό η ε, κυρία Σίπελ, παρακαλώ, ο καθένα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύσκολο αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι μας έχουμε να υποβάλουμε πολλές ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα προσπαθήσω να εστιάσω σε δύο-τρία θέματα. Μόλις διάβασα ε, ένα μια δημοσίευση στον τύπο από του υπουργού εσωτερικών υποθέσεων όπου γίνεται λόγο για προαιρετική επιστροφή ανθρώπων προ τη Λιβύη και τον Ήγηρα. Μήπω μπορείτε να μα πείτε τι ακριβώ γνωρίζετε από αυτού. Ε, είναι οι χώρες προέλευση των ανθρώπων που παραμένουν ε, στη Λιβύη, που πήγαν στη Λιβύη για να εργαστούν και τώρα κατά κάποιον τρόπο είναι παγιδευμένοι. Και αν γνωρίζουμε ότι έχουν άλλη χώρα προέλευση, πρέπει να κάνουμε ακριβώ έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο να επιστρέψουν στις πατρίδες τους αλλά να έχουν και μία προοπτική ε, για να μην έχουν και πάλι λόγο να εγκαταλείψουν αυτή την πατρίδα τους και να πάνε και πάλι ε, αναζητώντας ε, μια ασφαλή χώρα. Τώρα, για τη Λιβύη άκουσα σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία για την ακτοφυλακή της Λιβύης. Γνωρίζουμε όμως όλοι μας ότι η ακτοφυλακή της Λιβύης είναι ένα είδος παραστερητικής ή υποστερητικής οργάνωσης. Δεν είναι ακριβώς ακριβώς οι ίδιοι υπάλληλοι του Δημοσίου. Μπορείτε να μας ενημερώσετε λιγάκι για αυτούς ε, αυτοί που εργάζονται για την ακτοφυλακή της Λιβύης ισχύει ότι είναι και οργανωμένοι με οργανωμένο έγκλημα και εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους ε, που παγιδεύονται στην Λιβύη και τους ε, ξαναγκάζουν σε εργασία, τους αντιμετωπίζουν ως ένα είδος δούλους. Όσον αφορά τώρα την επανεγκατάσταση από περιοχές ε, που μένονται οι συγκρούσεις, ε, ε, τι θα γίνει τελικά με τα κράτη-μέλη που δεν τάσσονται ιδιαίτερα υπέρ της επανεγκατάστασης και κάποιες ερωτήσεις για την ασφάλεια. Μιλήσατε για την ρίζοσπαστικοποίηση και την αντιμετώπιση της. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε επίσης για ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο που θα ασχολείται με αυτό αυτό ακριβώς το θέμα. Ελέγχετε κάποια άποψη συγκεκριμένη για το τι ακριβώς διαδραματίζεται στα κράτη-μέλη και πώς ένα τέτοιο ευρωπαϊκό κέντρο θα μπορούσε να ενταρρύνει τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν περισσότερο με αυτά τα θέματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η ε, τρομοκρατία. Η κυρία Γκόμες, παρακαλώ, επόμενη. Ευχαριστώ πολύ για τη Λιβύη. ο πρέσβης κ. Κόμπλερ που ήταν ο ειδικό εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Λιβύα μέχρι τον, το τέλος Ιουνίου, ήταν ο Γερμανός πρέσβης συγκεκριμένα, ε, ήρθε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πριν από τρεις εβδομάδε και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει στρατόπεδα συγκέντρωσης, έτσι τα ονόμασε, γιατί πράγματι ε, λαμβάνουν χώρα τρομακτικά βασανιστήρια, ε, χωρίς να υπάρχει καμία εξωτερική παρακολούθηση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η να το πούμε έτσι, ε, ε, ε, βασίζονται στο, στην ύπατη αρμοστία του για τους πρόσφυγες, η οποία όμως δεν έχει σχεδόν καθόλου τοπική παρουσία, επιτόπου παρουσία. υπάρχουν ε, ελάχιστοι εκπρόσωποι της ΑΚΝΟΥΡ, του, λίγοι του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης τι γίνεται έτσι ώστε να μην πληρώνουμε με δικά μας χρήματα τη δημιουργία και τη λειτουργία στα στρατοπέδων συγκέντρωση βασανιστήριων κλπ. Εγώ το 2011 και 2012 είχα επισκεφθεί μερικά τέτοια και έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρη ότι είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα, μετά, πώς παρακολουθούμε την κατάσταση έτσι ώστε η εκπαίδευση ε, της ακτοφυλακής της Λιβύης ε, λειτουργεί και δεν μας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Διότι ακούω ότι έχουν γίνει πυροβολισμοί εναντίον Ιταλικών σκαφών και μετά ζητούσαν συγγνώμη επειδή νόμιζαν ότι ήταν μετανάστες. Δηλαδή ήταν μετανάστε θα ήταν εντάξει να του πυροβολήσουν. Πώς μπορεί να συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την πολιτική αν δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Μία μόνο ερώτηση για την πέμπτη οδηγία ε, κατά του, της νομοποίησης παρανόμων προσόδων. Ελπίζουμε ότι η Προεδρία θα Λήξη με αυτό το θέμα διότι είχε μπερδευτεί το θέμα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Προεδρίας. Θα ήθελα να σα ζητήσω να προχωρήσουμε με αυτό το φάκελο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Ευχαριστώ. Η μηνοποίηση παρανόμων εσόδων είναι αύριο με τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Η Μπιόρκ. Ευχαριστώ τον ε, Υπουργό και για την ε, έκθεση την οποία συνεργαστήκαμε για την ε, επανεγκατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας. Να προσθέσω στις ερωτήσεις κυρία Σίπελ. Στην δήλωση της 6 Ιουλίου στο ανακοινωθέν τύπου λέτε ότι θα αυξηθούν οι επανεγκαταστάσεις από περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις, πολεμικές συγκρούσεις. Ε, τι, αυτό είναι ευρωπαϊκό η πρωτοβουλία. Εθνική πρωτοβουλία θα είναι σύμφωνα με την, ε, κάτι παρόμοιο με τη συμφωνία με την Τουρκία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγο περισσότερε πληροφορίες γι' αυτό. Δεύτερον, ε, για το Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Είχαμε ορισμένοι ευρωβουλευτέ από διάφορε πολιτικέ ομάδε στείλει μια επιστολή, εκφράζαμε τι ανησυχίε μα. Και ποιε ήταν αυτέ. Μία είχε σχέση με τον δεοντολογικό κώδικα ορισμένων ε, μη κυβερνητικών ανανώσεων προβαίνουν σε διασώσεις. Ε, δεν είναι σωστό να κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι σώζουν ζωές. Ε, εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ευρωπαϊκή δραστηριότητα ε, διάσωσης, ε, ε, οπότε δεν κάνουμε το καθήκον μας. Αν περιορίσουμε και τις αντίστοιχε δραστηριότητε των μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα χάσουμε και άλλες ζωές και θα έχουμε την ευθύνη. Και σωστά θα έχουμε την ευθύνη και θα μας βαρύνει ε, το κρίμα. Μετά, οι συνάδελφοι ε, αναφέρθηκαν στην ε, υποστήριξη στην ε, δίθεν λιβιαϊκή ακτοφυλακή. Από ό,τι λέει ο ΕΕΠΡΟΚΤΕ, πρόκειται για παραστατευτικές οργανώσεις προβαίνουν σε ε, ολέθρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η συνεργασία με την λεγόμενη Λιβιακή ακτοφυλακή μου φαίνεται ότι είναι εκτός ορίων. Τέλος, να πω κάτι για τις ευθύνες μας για το μέλλον. Νομίζω ότι η ακρογωνία λύθη για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης δεν είναι τα σύνορα και οι επιστροφές, αλλά η αλληλεγγύη και ο καταμερισμός ευθυνών. Και θα πρέπει να τα καταφέρουμε και το Συμβούλιο θα πρέπει να τα καταφέρει εμείς. Εργαζόμαστε σκληρά και βασιζόμαστε σε εσά να κάνετε το ίδιο να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ε, πρέπει να σας πω ότι είναι χαρά για μένα που μου δίνετε ευκαιρία να σας ξανασυναντήσω. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε και για αυτά που ε, παρουσιάσετε ως προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Εγώ θα εστιάσω σε δύο θέματα. Στη νέα υπηρεσία για το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο σύστημα Schengen. Όσον αφορά αυτή τη νέα υπηρεσία, το νέο γραφείο, ε, χαίρομαι που είπατε ότι είσαστε αποφασισμένοι να το ολοκληρώσετε το θέμα, να το κλείσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πράγματι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό οργανισμό για τη χορήγηση ασύλου και αυτό το χρειαζόμαστε γρήγορα. Όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Schengen, χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Ε, πιστεύω ότι είναι προτεραιότητα για σας ε, και αργότερα, σήμερα το απόγευμα, θα ακούσουμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει και αυτό να κάνει κάτι γρήγορα. Το σύστημα SIS ε, είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των πολιτών μας ήδη τώρα, άρα δηλαδή θα πρέπει να καταλήξουμε το στεμό των δυνατών σε πολιτική συμφωνία και προσβλέπω στη δική σας υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Έλλη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι τα καλύτερα για την Προεδρία σας. Ε, βεβαίως ξεκινάτε με πολύ δυσάρεστες συνθήκες. Είναι ε, τελείως τρελό το ότι το Συμβουλίο ξέχασε τις δεσμεύσεις του σχετικά με τη μετεγκατάσταση και το θέμα του Δουβλίνου. Και προσπαθούν να ξεφύγουν από την αλληλεγγύη και ούτε καν και στο Συμβούλιο δεν συζητήθηκε αυτή η πρόταση που έγινε από την Επιτροπή. Θα ήθελα να σας ε, ερωτήσω, επειδή είπατε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ στο θέμα τη συνθήκη του Βλήνου. Μήπω μπορείτε λιγάκι να διευκρινίσετε. Εγώ το βρίσκω ντροπιαστικό το ότι το Συμβούλιο συμφωνεί μόνο στο να σε εξωτερικούς παράγοντε τα θέματα των ε, συνόρων μα. Το πρόγραμμα δράση εστιάζεται ακριβώ σε αυτό τη εξωτερική ανάθεση εστιάζεται στην ε, μετεγκατάσταση, στην επαναπρόθεση. Ε, μην ξεχνάτε ότι στι λιβικέ ακτέ η ακτοφυλακή του φεκίζει τους μετανάστες την Πέμπτη πήγα στην Κατάνια και επισκέπτηκα ένα από αυτά τα σκάφη ε, της SOS ε, Μεσόγειος, της SOS Μεντιτρανέ και μας ε, είπαν και το είδαμε κιόλας ότι πολλά από αυτά τα άτομα έχουν εμφανεί τα σημάδια από τα βασανιστήρια που υπέστησαν στη Λιβύη. Και τι κάνει η Ευρώπη, προσπαθεί να τους κρατήσει εκεί που είναι, σε μια χώρα όπου ποδοπατιούνται καθημερινά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα δηλαδή είναι η ΜΚΟ, το αποδιοπομπαίος τράγος είναι σαν αυτές να φταίνε και όχι ότι φταίει το ότι δεν υπάρχει μια σωστή ευρωπαϊκή απάντηση έτσι ώστε να υπάρχει και ασφαλής πρόσβαση σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η μόνη λύση για να υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και για να αποφύγουμε μόνο ορισμένα κράτη όπως η Ιταλία και η Ελλάδα να είναι το μόνο σημείο πρόσβασης αν θέλει κανείς να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ράντεφ, παρακαλούμε. γαλλικά έχει. Ιταλικά. Κανένα δεν έχει. Χάλασε και το μικρόφωνο. Ναι. Τι έχει η ομάδα, ποιος έχει την ομάδα. Δεν έχουμε. Είχαμε, είχαμε την έφερε τότε. Τι γλώσσα είναι αυτή που μιλάει αυτός. Αφού δεν... Το μικρόφωνο σου δεν ξέρω. Sorry, colleagues, we're just checking that. Oh, Συναδελφοί, ε, υπάρχει ένα, τεχνικής, ε, ένα τεχνικό πρόβλημα. Να μιλήσουν πρώτα οι άλλοι και μετά να επανέλθετε εσείς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο ομιλητή, στην ομιλήτρια από την Εστονία ε, ελπίζω να έχουμε μετάφραση από τα αισθανικά, να μπορώ και εγώ να μιλήσω σήμερα εστονικά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ερωτήσω το εξής. Είπατε ότι η Εστονία ε, θα, ήθελα, θα ήθελε να ε, προχωρήσει με την επεξεργασία των δεδομένων, ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές υποθέσεις. Κατά την άποψή σας, Ποιε είναι οι δυνατότητε που υπάρχουν έτσι ώστε να ε, επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχου των μεταναστών. Φοβάμαι ότι οι μετανάστε ε, παραμένουν στου καταβλισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί καθυστερεί όλη αυτή η διαδικασία. Και είπατε μετά ότι η προστασία των δεδομένων είναι προτεραιότητα, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω το εξή. Τώρα, υπάρχει και λιγότερο από ένα χρόνο για να εφαρμόσετε αυτό ο κανονισμό περί τη προστασία δεδομένων. Υπάρχει όμω ένα κανονισμό ε, για την ιδιωτική σφαίρα ε, που θα εφαρμοστεί και αυτό σύντομα. Πάμε από τα δύο δηλαδή. Εσείς τι ακριβώ προβλέπετε, πώς θα δουλέψει το Συμβούλιο ώστε να έχουν γίνει όλα όσα είναι απαραίτητα μέχρι το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς. Κύριος Λέναρς και μετά θα επανέλθω στον κύριο Ράντεβ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστούμε που ήρθατε. Νομίζω πράγματι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε κατά τους επόμενους μήνες στο, στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και προσβλέπω στη συνεργασία. Και εγώ δύο ερωτήματα σύντομα. Το ένα αφορά τη διαλειτουργικότητα. Είμαι ακράδοτα πεπισμένος ότι η διαλειτουργικότητα είναι μία από τις, ε, θα είναι μία από τις προτεραιότητες στους επόμενους μήνες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ανησυχίες και υπάρχει και ένταση. Μερικοί λένε να πάμε πιο πολύ στην διαλειτουργικότητα και να είναι πιο ισχυρή η προστασία της ιδιωτικής εσφαίρα. Τώρα πώς τα βλέπετε εσείς ακριβώς όλα αυτά. Πώς προτίθεστε να εργαστείτε από αυτόν κατά τους επόμενους έξι μήνες δεύτερη μου ερώτηση αφορά την ε, μετανάστευση και τη χορήγηση ασύλου. Ε, ένας βασικός, ένα βασικό στοιχείο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα είναι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας επαναπρόθεσης ε, των προσφύγων και μεταναστών. Δουλεύουμε με το Eurodac, με το σύστημα SIS. Έχετε καμιά άλλη ιδέα για τους επόμενους έξι μήνες, κάτι άλλο που μπορεί να γίνει, έτσι ώστε η πολιτική επιστροφή των ανθρώπων να είναι πιο αποτελεσματική. Είσαστε έτοιμος τώρα, είμαστε εντάξει, μπορεί να ε, μιλήσει ο κύριος Ράντεφ. Ναι, πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, μία από τις ε, μεγαλύτερες ε, προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεταναστευτικό. Μιλάμε γι' αυτό εδώ και πολύ καιρό η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιταλία, παραμεθόριες χώρες αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση ακριβώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Και μιλάμε εδώ και αρκετό καιρό για την ανάγκη ότι πρέπει να τροποποιηθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου, κυρίως η διαδικασία υποδοχής των μεταναστών. Η Ιταλία τώρα επιβεβαιώνει ότι χρειαζόμαστε ε, ταχύτερα και πιο μακροπρόθεσμα μέτρα για να μπορούμε να υποδεχτούμε τους μετανάστες στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση να κάνετε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε ε, να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου. Οι χώρες προέλευσης και οι χώρες διέλευσης ε, θα πιστούν ότι, αν γίνουν όλα αυτά, θα πιστούν ότι νιώθουμε αλληλέγγυοι εναντί τους. Και αυτά βέβαια θα πρέπει να συμβαδίζουν και με τη διαδικασία επαναπροώθηση των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα νομικό αίρισμα να παραμένουν εδώ και αυτοί πρέπει να επιστραφούν το στομότερο δυνατόν στις χώρες προέλευσής τους ή διέλευσης. Ελπίζω λοιπόν ότι θα περιοριστεί, όπως σας είπα, το χρονικό διάστημα από την ώρα που απορρίπτεται μια της χωρίς ασύλου μέχρι να επιστρέψει ο άνθρωπος αυτός ε, στη χώρα ε, προέλευσης του. Επόμενος ομιλητής ο κύριος ε, Βόιτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, είπατε πολύ σωστά ότι έχουμε την υποχρέωση να ε, προστατεύουμε τους ε, πολίτες μας. Από αυτό το Σαββατοκυριακό γνωρίζουμε όμως ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να ε, λάβει χώρα σε όλες τις χώρες. Η, τώρα τι έγινε στο Αμβούργο, 20.000 αστυνομικοί μπόρεσαν να προστατεύσουν την συνάντηση κορυφή, όχι όμως τους πολίτες του Αμβούργου. Και είπατε επίσης ότι θα πρέπει μεταβατικά και κατά περίπτωση να επανεισάγονται κάποια μέτρα. Δηλαδή τι εννοείται, συνοριακή έλεγχη, να υπάρχει και μία τράπεζα δεδομένων για ακροαριστερούς εξτρεμιστές και στο μέλλον να μπορεί κανείς να προλάβει ε, την έκρηξη βίας και όχι να προσπαθεί να την ε, θεραπεύσει και να την αποκαταστήσει εκ των υστέρων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για τις ε, ερωτήσεις σας και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Υπουργό ε, να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Συγγνώμη, ήθελαν και άλλοι να πάρουν το λόγο, εγώ αυτά τα ονόματα είχα. Νόμιζα ότι είχατε σημειώσει την επιθυμία μου Ε, να μιλήσουν και πράσινοι. Η γλώσσα σώματό μου δεν είναι και τόσο συγκρατημένη. Ποτέ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, εντάξει, ε, συντομία, Πρόεδρε. Η συζήτηση των τελευταίων ε, δύο εβδομάδων αφορά την τεράστια εισρωή μεταναστών και προσφύγων στην Ιταλία. Και η ανταπόκριση που είδαμε κοινή αντίδραση Γαλλίας, Ιταλίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εστιάζει ιδιαίτερα στις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα σκάφη των ΜΚΟ που ε, διασώζουν πρόσφυγες και μετανάστες κοντά στα σύνορα τι θα είναι αυτός ο κώδικας για τις ΜΚΟ και τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να πετυχάνεται ο στόχος μέσω αυτού του κώδικα και κατά πόσο θα πρέπει να επηρεάζονται ε, και τα εμπορικά σκάφη ε, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Προβλέπετε ότι θα υπάρχουν ασφαλείς λιμένες ε, κοντά στην περιοχή πέραν της Ιταλίας, στο εγγύηση σε μέλλον. Υπάρχει μια συζήτηση για την Τινησία, αλλά από την έκθεση που λάβαμε, για μια συζήτηση που δεν θα γίνει σήμερα για την επανεσδοχή, η συμφωνία με την Τινησία, ουσιαστικά, οι διαπραγματεύσεις μάλλον δεν προχωρούν ουσιαστικά. Ποια είναι η θέση λοιπόν της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε αυτό το θέμα. Με την κατάσταση. Έχουμε Ιούλιο το Σεπτέμβριο. Κλείνουν τα δύο έτη όπου ε, τα δύο έτη δηλαδή συμπληρώνονται του προγράμματος μετακατάστασης όλων αυτών των ανθρώπων που βεβαίως και δεν επιτυγχάνεται τελικά ούτε κατά διάνοια. Τι προβλέπετε ότι θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο. Και τέλος, για τη διαλειτουργικότητα, Πρόεδρε, η ομάδα μου ε, προσπαθεί να καταλήξει σε μία άποψη. Θα θέλαμε κάπως να κατανοήσουμε αν προβλέπετε αυτόματες και υποχρεωτικές ανταλλαγές πληροφοριών ή αν υπάρχει ακόμα δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να πούν όχι, εμείς δεν θα ε, μεταφέρουμε και δεν θα ανταλλάζουμε με τους πάντες ε, δεδομένα αυτομάτως εντός της Ένωσης βεβαίως. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, που δεν σας έδωσε το λόγο πριν. Η Μπάρμπαρα και άλλοι συνάδελφοι θα μιλήσουν στο επόμενο θέμα, να τους ευχαριστήσω και την υπομονή τους, γιατί ε, λίγο θα καθυστερήσουμε. Εν συντομία να πω ότι έχουμε εδώ και αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Εστερικών της ε, Βουλγαρίας. Τους οποίους συνοδεύει ο κ. Ράντρεφ, νομίζω, εδώ. Καλώς ήρθατε στη συνεδρία της Επιτροπής μας. Και οι Βούλγαροι συνάδελφοι εργάζονται ε, για να προετοιμάσουν την επόμενη Προεδρία. Υπουργέ, τώρα μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς από εσά που σας έχω ήδη συναντήσει και προσωπικά, ε, καθώς ήσασταν ε, εισηγητές, ισκιώδεις εισηγητές, για πολλές σημαντικές προτάσεις. Και αυτό με έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να κατανοήσω τον τρόπο λειτουργίας ε, του Επινοβουλίου τις προτεραιότητες και τις ταχύτητες με τις οποίες εργάζεστε εδώ. Τα ερωτήματά σας θα τα ε, μοιράσω σε τρεις ε, ξεχωριστές κατηγορίες. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω βέβαια ε, ανακατηγορία τις παρατηρήσεις μου για να παρουσιάσω έτσι και το όραμα της ε, Προεδρίας μας και πώς ε, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Πρώτα απ' όλα περνάω στο πλέον σημαντικό ζήτημα, κυρία Σίπελ και Πολλοί άλλοι συνάδελφοι το έθιξαν, δεν θα τους κατανομάσω όλους, για το σχέδιο δράσης στην Ιταλία και μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Πρώτα απ' όλα, η Ιταλία ήρθε σε επαφή με την Εστονία πριν από 10 ημέρες, λίγες μέρες δηλαδή πριν από την άτυπη συνάντησή μας και μας ε, ζήτησε η Ιταλία να συμπεριλάβουμε αυτό το σημείο στη μέσα διάταξη. Εμείς ανταποκριθήκαμε πολύ γρήγορα. Λίγες μέρες μετά Είχαμε την κοινή συζήτηση Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Παρίσι. Οπότε γνωρίζαμε ε, το περιεχόμενο σαφώς ε, των συζητήσεων αυτών. Ήδη λοιπόν ξέραμε ότι θα υπήρχε αυτό το ζήτημα ε, του σχεδίου δράση για την Ιταλία ως ε, πρώτο και πιο σημαντικό σημείο μέσα στη διάταξη του Ταλίν. Κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι δεν μπορούσαμε εκείνη τη στιγμή να υιοθετήσουμε επίσημες ε, αποφάσεις γιατί είμαστε σε ένα άτυπο συμβούλιο. Είπαμε όμω ότι χαιρετίζουμε το σχέδιο δράσης. Και Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις εκεί, σε αυτό το κείμενο. Και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι όντω ε, ακαθόδε το ζήτημα, υπήρξαν μακροσκελεί συζητήσει και είναι πραγματικά ένα σχέδιο δράσης για την ε, Ιταλία και τις ΜΚΙΟ. Και βεβαίω θα θέλαμε να δούμε και τη συνεισφορά των υπόλοιπων κρατών μελών. Επομένω, θα διοργανώσουμε συναντήσει σε διάφορε ομάδε εργασία για αυτό το σχέδιο δράση και ελπίζουμε εκεί να συμβάλλουν και όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα συντονίσουμε τη συνεργασία μας με τις ΜΚΟ, όχι για να τις περιορίσουμε. Προσπαθούμε να συντονίσουμε την συνεργασία μας. Ένα παράδειγμα που έδωσε και στο Ταλίν. Αν έχουμε έναν ε, πυροσβέστη, τέλο πάντων και την πυροσβεστική με του επαγγελματίε και του εθελοντέ, τότε πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, δύο. Αλλιώ χαθήκαμε. Και εδώ τον ίδιο στόχο έχουμε λοιπόν, συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ που πραγματικά σώζουν ζωές στη θάλασσα, έτσι. Και φυσικά και δεν θα τις πιέσουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούν πλέον να επιτελέσουν το έργο τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για την άτυπη συνάντηση δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία τέτοια συζήτηση. Τώρα για το θέμα της Λιβύης. Για την ε, λιβυκή Εκτοφυλακή. Και το θέμα των πολιτικών δυνάμεων. Εδώ έχουμε ορισμένες εμβολίες, όμως ε, πρέπει ε, κάπως να έχουμε στο πλευρό μας τη Λιβύη, είτε μας αρέσει είτε όχι. Οπότε δεν μιλούμε για τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο, αλλά και το, ε, τα λιβικά σύνορα προς τον Νότο. Γιατί από εκεί έρχονται ε, πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Μία από τις μεγαλύτερες ροές ε, έρχεται από τον Μπαγκλαντές διασχίζουν ε, την έρημο και πολλοί μάλιστα χάνουν και τη ζωή τους εκεί. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία πραγματική ευκαιρία να βάλουμε τέλος ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεργασία με τη Λιβύη. Έχουμε και το ε, καταπίστευμα για την Αφρική, το οποίο έχει θεσπιστεί. Σίγουρα θα χρειαστεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τα κρατημέλη προκειμένου να ε, προχωρήσει. Θέλουμε καλύτερη συνεργασία με αυτούς που βρίσκονται ήδη εκεί. Χρειαζόμαστε κατάρτιση και μόνο και μόνο κατάρτιση θα χρειαστεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Προχωρώ τώρα στην αλληλεγγύη. και αυτό μας συνδέει και πάλι με το θέμα του Ταλίν και εδώ πρέπει να το μοιράσουμε σε δύο ζητήματα. Το θέμα της Ιταλίας προέκυψε ε, μάλλον ε, απρόσμενα. Ε, στη δεύτερη μέρα συζητήσαμε λοιπόν ε, την αλληλεγγύη, τη μεταρρύθμιση του ε, κανονισμού ε, του Δουβλίνου και το θέμα της ευθύνης. Πρέπει να τα δούμε από κοινού αυτά τα πράγματα. Ίσως μακροπρόθεσμα να πρέπει να τα, διαχειρι... να τα διαχωρίσουμε. Αλλά το θέμα της Ιταλίας μας έδειξε ότι πρέπει γρήγορα ε, να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια. Ο κανονισμός του Δουβλίνου μπορεί να αποτελέσει τη βάση όλων αυτών των ενεργειών. Ξέρουμε ότι όλα αυτά τα θέματα που αφορούν ε, την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου βρίσκονται προ το τέλο των συζητήσεων, οπότε πρέπει να είμαστε πάνω κάτω έτοιμοι, προχωρώντα προς τους τριμερεί διαλόγου. Το πιο σημαντικό θέμα βέβαια είναι η αλληλεγγύη. Και σίγουρα εκεί που θα κολλήσουν τα πράγματα είναι το γεγονό ότι, στα... οι απόψει δίστανται σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη στη... μεταξύ... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζητήματα γιατί σαφώς και υπάρχει εθνική κυριαρχία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μια πολύ αποτελεσματική πολιτική επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν ε, ισχυρή προστασία των εξωτερικών συνόρων, θα μας δώσει μια καλύτερη εντολή για να προχωρήσουμε. Οπότε τα κάτι μέλη που δεν βλέπουν ε, την αλληλεγγύη με τον ίδιο τρόπο που βλέπουν τα υπόλοιπα κρατη μέλη που θέλουν να συνεργαστούν, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εφαρμόσει τα δικά τη μέτρα προ αυτά τα κρατη μέλη, αυτό είναι η δική τη απόφαση, θα δούμε ποιες θα είναι αυτές οι αποφάσεις και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ βέβαια θα είχα την επιθυμία να εργαστούν από κοινού και επί μια βάση αλληλεγγύη όλα τα κρατημέλη. Αυτό θα προσπαθήσουμε μέσα στου επόμενου μήνε, γιατί θα θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση για αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου είναι κάτι αναπόφευκτο. Ε, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αυτή η κρίση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ιταλία θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και πιο βόρεια. Λοιπόν, θα περάσω τώρα σε ένα σημαντικό θέμα για την Εστονία, τη διαλειτουργικότητα. Πρώτα απ' όλα, τον 21ο αιώνα αυτή είναι η πραγματική μοναδική δυνατότητα που έχουμε για να ε, έχουμε πρόοδο ό,τι αφορά την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Άρα οι αρχέ επιβολή του νόμου πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν με έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό διασφαλίζεται μόνο όταν έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό ε, και διαλειτουργικό μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών υπήρχαν πολλά ζητήματα για την προστασία των δεδομένων. Και μπορώ να επιβεβαιώσω βάσει του εστονικού παραδείγματο ότι αν έχουμε πολύ καλά οργανωμένε βάσει δεδομένων, ε, αυτό μας επιτρέπει να ελέγχουμε καλύτερα αυτές, αυτές τις βάσεις και μπορούμε και πολύ πιο εύκολα να εντοπίσουμε τυχόν καταχρήσεις. μπορούμε να έχουμε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για τις ε, αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου οι πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα ε, να τυχάνουν χάνουν στις καλύτερες δυνατές προστασίας. Και αυτό διασφαλίζεται μέσω της χρήσης σύγχρονων διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων, που λειτουργούν πολύ καλύτερα από τις ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, γιατί τότε χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δουλειά για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, για το ΕΑΖΟ. Ε, το ανέφεραν οι συνάδελφοι. Πράγματι, αυτό το, φα... το φθινόπωρο θέλουμε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Σύστημα ανταλλήλωση προφοριών Σέγγεν. Από ό,τι ξέρω, Προχωράμε και εδώ, κυρίως στο φθινόπωρο θα υπάρξει πρόοδος. Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα εισόδου-εξόδου και για το αίτιας. Ήδη βρισκόμαστε πυλών σε ό,τι αφορά τις, ε, τους τριμερείς διαλόγους. Είμαστε κοντά λοιπόν σε μια συμφωνία και στο αίτια θα προχωρήσουμε σε τερμερίες διαλόγους στο φθινόπωρο. Για την ριζοσπαστικοποίηση και το Ευρωπαϊκό Κέντρο νομίζω ότι αυτό είναι μια μελλοντοστραφής ε, προσέγγιση την οποία και στηρίζω. Θεσπίστηκε βάσει όμως της εφιστάμενης αστυνομικής συνεργασίας, όπου ήδη υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, για ιστοτόπους που στηρίζουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Εγώ πήγα με τον ε, Επίτροπο Αβραμόπουλο στη Silicon Valley, όπου ε, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των μεγαλύτερων εταιριών δικτύων, μέσων κοινωνική δικτύωση που είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί μα. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε υπόψη ότι αυτές οι επιχειρήσει ανταγωνίζονται η μία την άλλη, παρόλα αυτά συνεργάζονται μαζί μα για να κατεβούν από το δίκτυο αυτά τα site ρίζους Βέβαια είναι πιο εύκολο για αυτές να συνεργαστούν με έναν συγκεκριμένο φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια, αν υπάρχουν και συγκεκριμένα κράτη-μέλη που θέλουν να συνεργαστούν με αυτέ τι εταιρείε στο πλαίσιο συγκεκριμένων υποθέσεων, μπορούν να το κάνουν. Αλλά τώρα εμεί μιλάμε γενικότερα για το θέμα τη απορριζοσπαστικοποίηση και τα μέτρα που λαμβάνουμε σε αυτό το τομέα. Τώρα, ένα ερώτημα που αφορούσε την μετεγκατάσταση, την επανεγκατάσταση μάλλον από τρίτες χώρες. Ως ε, Προεδρία καλούμαστε να ζητήσουμε από τα κάτι μελη ε, να επιτρέψουν ε, την ε, επανεγκατάσταση. Η Εστονία βρίσκεται κάπου στη μέση της κατάταξης σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα επανακατάστασης. Θα θέλαμε όμως να έρθουμε σε συμφωνία με την Ιταλία, γιατί για μας είναι σημαντικό οι συνεντεύξεις να γίνονται στην Ιταλία, εκεί στα κέντρα υποδοχή και μετά να γίνεται η ε, μετακατάσταση. Λυπάμαι αν έχω ξεχάσει κάτι, ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Και βέβαια ελπίζω ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον βέβαια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Οπότε ε, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία με του επόμενου μήνες. Και σίγουρα θα τα πω με πολλούς από εσάς ε, και θα μάθω και ποιε είναι οι δικέ σα προσδοκίε για αυτά τα ζητήματα κρίσης αλλά και τα ε, μακροπρόθεσμα πολιτικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ πολλά από αυτά τα θέματα μεταξύ αυτών και η Λιβύη είναι θέματα τα οποία εξελίσσονται, εκτιλίσσονται αυτή τη στιγμή, οπότε θα σας ξαναδούμε σύντομα. Στις 24 Ιουλίου θα λάβει χώρα το Συμβουλίο Υπουργών που θα εξετάσει το θέμα της Λιβύης. Και φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσετε για, για την έκβαση. Είναι τόσο πολλά τα θέματα που τρέχουν βέβαια που θα είμαστε όσο πιο ελαστικοί γίνεται σε ό,τι αφορά τις ε, ε, παρεμβάσεις σας εδώ και το, τη λογοδοσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα περιμένουμε και τον συναλληφό σας Υπουργό για ε, αρμόδιο θέματα δικαιοσύνης μεταξύ άλλων να μας μιλήσει και για το θέμα της νομοποίησης παράνομων προσόδων. Έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Θα περάσω λοιπόν στο επόμενο θέμα, σημείο 4. τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018, για τον κύριο Γέζεκ. Στο συγγνώμη που καθυστερήσαμε κύριε Γέζεκ, θα σας δώσουμε το λόγο. Είστε ο εισηγητής ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω θα τελειώσουμε πριν τις σκέμιση, γιατί ε, θα πρέπει να ε, φύγω. Στο τμήμα 3 του προπολισμού 2018 ε, οι διασμένες πληρωμών έχουν μειωθεί κατά 17,9% και 21,7% ε, οι ε, δεσμεύσεις πιστώσεων σε σχέση με το 2017. Ε, ή το όργανο ευελιξίας ε, είναι καλό, πολύ καλό που χρησιμοποιείται γιατί ε, προσθέτει 817 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι επαρκές για να αντιμετωπίσουμε τις διαρκώς ευκαιρόμενες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας, εδώ ο προϋπολογισμός μειώνεται κατά 35,6% σε σχέση με το 2017. Έχουμε πολλές ανησυχίες, κοινέ ανησυχίες ασφάλειας στην Ευρώπη και δεδομένου ότι μπορεί πολλοί ε, μαχητές ε, να επιστρέψουν από τη Συρία και το Ιράκ στο μέλλον, δεδομένου ότι το, ο, Ισλαμικό, το κράτος ε, χάνει μάχες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει απαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσει αυτή την αυξανόμενη απειλή. Με την ε, δημιουργία ενός σαφούς συστήματος εισόδου και εξόδου ε, θα πρέπει να έχουμε αρκετούς πόρους για να τα εφαρμόσουμε αυτά τα συστήματα. Αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το, το Ταμείο ε, ΑΜΙΦ ε, για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη βλέπει τις πόρους του να μειώνονται. Αντίθετα, η ε, η κάλυψη του αυξάνεται περισσότερο. Ε, εκτός από τη Βαλτική θάλασσα βλέπουμε στην ε, κεντρική Μεσόγειο να αυξάνονται οι ροές, κυρίως από τη Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την περίπτωση μιας ακόμα μαζικής εισόδου. Την τελευταία φορά ήμασταν τόσο πολύ λίγο προετοιμασμένοι σε δημοσιονομικά ε, που καταλήξαμε σε μια κατάσταση που χρειάστηκε μήνες για να την ελέγξουμε. Ε, οπότε μην ε, υποτιμούμε τις ανάγκες του Ταμείου ΑΜΙΦ για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη. Τέλος, να περάσω στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Είναι θετικό που η Κομισιόν πρότεινε αύξηση του προπολογισμού ε, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Όμως, ε, οι ανάγκες τους δεν καλύφθηκαν πλήρως. Το, η Ιουλίζα παίζει σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση αποτελεσματική ε, κατανομή πληροφοριών, διαμερισμό πληροφοριών και έχει λάβει και περισσότερες αρμοδιότητες ε, τελευταία. Αυτό λόγω χρειάζεται πολύ περισσότερους πόλους. Ε, η δράση μας στην τρομοκρατία, το οργανωμένο εμπόριο και την λαθρέα διακίνηση ε, έχουν αυξηθεί. Ε, οι δραστηριότητε εκεί και πρέπει να δούμε αν το προσωπικό αρκεί. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Ευχαριστώ budget headings Θα περάσουμε κατευθείαν στους κοιόδους συγητές και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Μπάρβαρα, εκ μέρους του ΕΛΚ. Καλωσορίζω αυτή ε, αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση του εισηγητή. Οι περικοπές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΑΜΙΦ και το ISF, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, είναι λυπηρές. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι περικοπές δεν δικαιολογούνται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μέτρα ε, ένταξης και ε, αποτελεσματικής επιστροφής. Ε, έχει καθυστερήσει η υιοθέτηση νομοθεσία και γι' αυτό λόγο ε, ε, ε Ορισμένοι υποστηρίζουν θα χρειάζεται λιγότερου λιγότερους πόρους η πολιτική ασύλου. όμω η Κομισιόν θα πρέπει σύμφωνα με τι υποσχέσει τη να υποβάλει ένα τροποποιητικό, μια τροποποιητική επιστολή μόλι ε, υιοθετηθεί η Σύμβαση του Δουβλίνου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση. Επίσης, χρηματοδότηση του ISF είναι απαραίτητη όχι μόνο για να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και να καταπολεμήσουμε το έγκλημα στον κυβέρνο χώρο, αλλά και για να καταπολεμήσουμε άλλου τύπου σοβαρά εγκλήματα διασυνοριακά, μεταξύ αυτών ε, δουλεμπόριο και ε, ε τρομοκρατία. Όλε οι υπηρεσίε σχετικέ με την δικαιοσύνη και τι εσωτερικέ υποθέσει θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώ, Συμφωνώ σε αυτό με τον Γενικό Συγητή. Γι' αυτό το λόγο η Eurojust, η Ulyssa και, όλοι, και όλες οι υπόλοιπε υπηρεσίες και οργανισμοί θα πρέπει να στηριχθούν. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε σαφώς στο κείμενο. Θα υποβάλουμε τροπολογίες σε ό,τι αφορά αυτήν και άλλες πτυχές και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε καλά με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. the shadow for the S&D Sylvie Guillaume, please. Σιλβί Κιγιόν για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Προς την ίδια κατεύθυνση θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και ο ίδιος και η κυρία Κουτρίσκα ε, εκφράζουν απογοήτευση ό,τι αφορά την δραστική μείωση των ε, ποσών στον τίτλο 3. Ο τίτλος 3 είχε βέβαια λάβει σημαντικά ποσά κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής κρίσης τα προηγούμενα χρόνια. Όμως αυτή η μείωση για το 2018 είναι πολύ γραφήρη, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπόψη το τι θα γίνει στους επόμενους μήνες. Δείτε τι συμβαίνει στην Ιταλία και στη Λιβύη. Τα ποσά τα οποία κατανέμονται στις διάφορες υπηρεσίες της αρμοδιότητας ε, ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, ιδιαίτερα στην ΕΑΣΟ, είναι ανεπαρκής, ανεπαρκή τα κεφάλαια, τα υπόρρια αυτή. Και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες που θα εκφράζουν τις ε, προτεραιότητές μας που είναι η υποδοχή και η ένταξη. Ευχαριστώ. Thank you very much, Sylvie. And there are no other shadows here. So... Δεν έχουμε άλλους και συγητές. Οπότε περνάμε στον κύριο Ντεπρί. Κύριος Ντεπρέ, λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με τις ε, κατευθύνσεις ε, του εισηγητή, του κύριου Γιάζεκ. Θέλω να τονίσω όμως δύο σημεία. Πρώτον, ε, κατόπιν της ψηφοφορίας που έγινε στην Επιτροπή, στη δική μας Επιτροπή, σε ό,τι αφορά το Eurodac. Κατόπιν αιτήματος της κυρίας Σιντβέλτ συμφωνήσαμε στην δημιουργία εντός της Europol μιας λειτουργικής ε, ομάδας, ενός λειτουργικού ε, τμήματος μάλλον, που θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί στενά τις ε, περιπτώσεις κατάχρησης ε, ε εις παιδιών και μη ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ήθελα να το υπενθυμίσω αυτό στον Πέτρ Γέζεκ. Χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό που να επιτρέψει τη Eurodac να φέρει σε πέρα αυτή την αποστολή που αποφασίσαμε να αναθέσουμε στην Eurodac. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τις, συναδέλφους που μίλησαν για το EU LISA, τον Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Μεγάλων ε, Συστημάτων Τεχνολογικής, Τεχνολογίας Πληροφορίας. Έχουν, ε, συντηρούν μεγάλες βάσεις δεδομένων στην EU LISA, πολύ σημαντικές βάσεις για την ασφάλεια αλλά και για την, ε, τα δικαιώματα τα προσωπικών δεδομένων κλπ. Το 2015 είχαν 2,5 εκατομμύρια ε, ε, προπολογισμό για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και το 2016 πέρασαν στα 6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ήταν ε, κακή η πολιτική αυτή. Πρώτα βάλουμε συγκεκριμένα κριτήρια προστασία δεδομένων και μετά αρνούμαστε να χρηματοδοτήσουμε επαρκώς τις δραστηριότητες αυτέ. Αυτά Συμφωνώ κατά τα άλλα με τον Πέτρ. Θα υποβάλουμε τροπολογίες μόνο για τα θέματα που οποία σας ανέφερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, αυτή ήταν και η άποψη του Συμβουλίου ε, που έλαβε χώρα την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν πίσω στον Πίτα για να κάνει σχόλια ε, σχετικά με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους και συζητητές για τη συνεισφορά τους και με μεγάλη μου χαρά να δεχτώ τις ε, τροπολογίες τους ε, που ε, θα αλλάξουν την πρόταση, όπως είπε προηγουμένως και ο Ζωρά. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ακούμε στα ακουστικά μας, κάτι δεν πάει καλά με τη μετάφραση. Λοιπόν, 20 Ιουλίου, καταλεκτική ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών και για τις ε, τροπολογίες για τον προπολογισμό. Επίσης, πολύ ωραία συνάδελφοι. Ε, ζητώ συγγνώμη για το επόμενο θέμα που ε, καθυστερήσαμε λίγο. Πάμε στο σημείο υπερθμών 5, Eurojust. Είναι ο προτινόμενος ε, νέος ε, κανονισμός που θα αντικαταστήσει την απόφαση του 2002 ε, για τη Eurojust 2013-0256 και νομίζω ότι ο στόχος ήταν η Κομισιόν να δώσει στη Eurojust μια νέα νομική βάση με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και Στόχος είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Eurojust, το Κοινοβούλιο ε, και τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες της Eurojust. Δεν θα πω τίποτα άλλο, έχουμε ήδη καθυστερήσει και Αξέλ να σου δώσω το λόγο. Ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Έχει το λόγο λοιπόν ο ε, συζητήτη να μα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τα διάφορα θέματα, ε, καταρχήν όσον αφορά ε, το πλαίσιο. Η Eurojust τα τελευταία χρόνια βοήθησε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και επίση και οι διαφορές ανάμεσα στα διάφορα νομικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γεβυρωθούν οι διαφορέ αυτές, να λύνονται γρήγορα τα νομικά προβλήματα και η Eurojust κατόρθωσε λοιπόν να ε, ικανοποιήσει αρκετά αιτήματα δικαστικής αρρωγής και με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατόν και να βελτιωθεί η υπερεθνική δίωξη. Από την άλλη πλευρά, τι γίνεται, διαπιστώνουμε ότι η διασυνοριακή εγκληματικότητα, η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, κυβερνοεγκληματικότητα, κυρίως η πορνογραφία για τα μικρά παιδιά. Αυτά όλα είναι αξιόπινες πράξεις οι οποίες περνάνε τα σύνορα και οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από ιδιαίτερα κινητικά άτομα άτομα που κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, αν θέλετε, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμεθα. Έτσι λοιπόν η Eurojust είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και για τον συντονισμό των αρμόδιων δικαστικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Είναι επίσης αρμόδια και για έρευνες που γίνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια σχετική πρόταση που αφορά στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία σε αξιόπινες πράξεις. Αυτό έγινε ήδη το 2013. Το Συμβούλιο το 2015 ε, όρισε την κατεύθυνση και όρισε και τις διατάξεις που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα επανέλθω σε αυτό. Αυτή η δική σχέση ανάμεσα στη Eurojust και την ε, Εισαγγελία και το γεγονός το γιατί υπήρξε καθυστέρηση νομίζω ότι ε, αυτό τελικά οδήγησε στο να μην προχωρήσουμε τόσο πολύ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο είχαμε κατά νου. Περίμενα λιγάκι σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης, ε, γιατί όλη αυτή η διαδικασία υπάγεται στην κανονική νομοθετική διαδικασία και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ε, φτιάχνει κομματάκια. Το Κοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθεί ε, συνολικά και μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν δυνατόν. Τώρα όμως υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις να επανέλθω και να πω κάτι. Η σχέση ανάμεσα στη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Συγκυλία, αυτό είναι το σημείο κλειδί. Και γι' αυτό λοιπόν αναγκαστήκαμε να περιμένουμε τόσο πολύ. Η διαδικασία αυτή με τη Eurojust, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους κοιόδης συζητήθηκε και όσον αφορά το σχέδιο της έκθεσης γενικότερα. Να πω το εξή. Εγώ ως εισηγητής τάσομαι υπέρ της άποψης του Συμβουλίου και θέλω να σας πω ότι ε, σημαντικά τμήματα της ε, έκθεσης ε, τα έχω προσαρμόσει στην κατεύθυνση που έχει ορίσει το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάλλου έχει ορίσει μέτρα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κατέστη απαραίτητη η μεταρρύθμιση της Eurojust, διότι στο άρθρο 86 της συνθήκης αναφέρεται ότι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας πρέπει να προκύψει από την Eurojust. Όσον αφορά όμως την ΕΠΟ, αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επ' αυτής ε, αρμόδια είναι 20 κράτη. Εν ε, βέβαια, ήταν 19 αλλά προσχώρησε και η Ιταλία και έγιναν 20. Και αυτά τα 20 ενδιαφέρονται να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία. Το να υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το θέλουμε όλοι μας, πόσο μάλλον εγώ. Βέβαια κάτω από την προϋπόθεση ότι ισχύει η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και επίσης ε, η δίωξη ε, θα εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα στα κράτη-μέλη. Η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει, όπως σας είπα, να προκύψει και το να υπάρχει εισαγγελία με βάση μια ομόφωνη απόφαση, αυτό θα προσέθεται υπεραξία στην δικαιοσύνη. Δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο. Ε, το προσπαθήσαμε, αλλά τώρα να ασκήσω και λιγάκι κριτική, δυστυχώς οι αρμοδιότητες πρέπει να επιμερίζονται ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη Eurojust και τα κράτη-μέλη. Βέβαια, οι αρμοδιότητες να ορίζονται με απόλυτη σαφήνεια, έτσι ώστε να μην προκύπτουν κενά, αλλά ούτε και επικαλύψεις. Όσον αφορά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για αξιόμενες αξιόπινες πράξεις που έχουν σχέση με οικονομική ζημιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επ' αυτού η Ευρωπαϊκή Αγγελία δεν έχει απόλυτη αλλά μερική αρμοδιότητα. Ε, ακριβώς λόγω αυτού θέλω να σε επισημάνω τη σύγκρουση συμφερόντων. Και θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα εντάξουμε στον ορισμό των αρμοδιοτήτων. Κατά την άποψή μου, και αυτό αναφέρεται στην έκθεση, η Eurojust ε, παραμένει αρμόδια για αξιόπινες πράξεις που έχουν σχέση με οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποτεδήποτε δεν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο έτσι ώστε να μην έχουμε κενά. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Eurojust εξακολουθεί να παραμένει αρμόδια για εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και Στόχο είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών για να αποκαλυφθεί η οικονομική ζημιά ει βάρος τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Ένα μεγάλο κομμάτι της έκθεσης αφορά την προστασία των δεδομένων. Και εδώ στηρίζω κυρίως τη διαφοροποίηση που έχει κάνει το Συμβούλιο ανάμεσα σε φυσικά άτομα, ε, μάλλον δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα άτομα και άλλα διοικητική φύσεως δεδομένα. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να ισχύουν οι διατάξεις εκείνες οι οποίες προβλέπονται για λειτουργικούς σκοπούς, ενώ η έκθεση της αδέλφου κυρίας Έρνστ του κανονισμού 54-2000 αφορά την θεσμική προστασία δεδομένων που έρει τα διοικητικά δεδομένα. Ως εκ τούτου χρειαζόμαστε αυτή τη διαφοροποίηση και στην έκθεση. Αυτοί οι ειδικοί κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων ισχύουν και για την Europol. Με βάση τον κανονισμό 2016 που έχουμε ήδη εγκρίνει και ο οποίος ε, κανονισμός θα ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο πλαίσιο του κείμενου κανονισμού ε, του 45-2001, ο κανονισμός αυτός δεν πρέπει να επεκτείνεται στα λειτουργικά δεδομένα. Όσον αφορά τώρα τη δομή και την οργάνωση της Eurojust, το Συμβούλιο είχε προτείνει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις ε, λειτουργικές και τις διοικητικές, ε, τα λειτουργικά και διοικητικά καθήκοντα. Εγώ υιοθέτησα αυτήν την προσέγγιση στην έκθεσή μου και στόχος είναι η Eurojust να, είναι, ε, να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά όπου η Eurojust ε, θα στηρίζεται από τα κράτη-μέλη μέσω του εκτελεστικού συμβουλίου. Άρα δηλαδή η Eurojust θα μπορεί να εστιάζει και να στοχεύει μόνο στις λειτουργικές διαδικασίες. Αυτό που δεν φύγω είναι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Εκτελεστική Επιτροπή. Εκεί προτάθηκαν δύο εκπρόσωποι της Κομισιόν. Εγώ λέω να υπάρχει μόνο ένας, γιατί και στην Europol ένας υπάρχει. Αυτό έχουμε προβλέψει. Και γι' αυτό και εγώ προσάρμοσα την έκθεσή μου. Ε, και κάτι άλλο που αφορά στο Brexit στην Ιρλανδία και στη Δανία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον ε, κανονισμό. Και η Δανία ε, δεν συμμετέχει, μέχρι τώρα δεν δεσμεύεται και αυτή η μη συμμετοχή αυτών των κρατών είναι κρίμα, διότι στην ε, ποινική και δικαστική συνεργασία χρειαζόμαστε όλα τα κράτη. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτήν την έκθεση προτείνω ε, με αυτά τα κράτη να συνάψουμε μία συμφωνία συνεργασίας και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και εμείς κύριε Βος, πάμε τώρα στους ε, σκιώδης ηγητές ε, και δίνω το λόγο στους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Κάουφμαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Φως, ο οποίος παρουσίαζε το θέμα του εκτενέστατα. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω που υπάρχει η δυνατότητα ε, να ασχοληθούμε με το κείμενο αυτό και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Και χαίρομαι που η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών έχει μετατεθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως όλοι σας γνωρίζετε, αυτή την εβδομάδα είμαστε μόνο στις Βρυξέλλες και επειδή το θέμα καθυστέρησε τόσο πολύ, ε, δεν θα ήταν δυνατόν και εμείς ε, να καταθέσουμε τις ε, τροπολογίες μας ε, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Φως επισήμανε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ήδη τεσσάρων ετών και εντωμεταξύ έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δηλαδή εντωμεταξύ έχουμε σχεδόν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ως εκ τούτου είναι σημαντικό και έτσι είχαμε συμφωνήσει, όταν θα είναι σαφές πώς θα εργάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τότε είχαμε πει ότι ασχοληθούμε με την αποκαλούμενη λισαβονοποίηση, συσσαγωγικά πάντα, της ε, Eurojust. Δηλαδή, να υπάρχει σαφή διαχωρισμός ε, εξουσιών, ε, να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Γιατί και οι δύο θεσμοί έχουν αρμοδιότητα ε, για συγκεκριμένα θέματα που τους έχουν να τεθεί. Ένα θέμα ε, θέλω να δείξω που νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη συγκεκριμένα. Εν τω μεταξύ έχει υπάρξει αξιολόγηση της Eurojust. Αυτό έγινε το 2015. Βέβαια τότε ίσχυαν άλλες ε, προϋποθέσεις. Πάντως ε, νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δούμε κατά πόσον από αυτή την αξιολόγηση η οποία έγινε μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής και η οποία, εντάξει και αυτή είναι δύο περίπου ετών, να δούμε λιγάκι κατά πόσον τώρα πράγματι τα έχουμε ε, συμπεριλάβει όλα αυτά που είπε ο κύριος Φως. Και κάτι τελευταίο, ε, σχετικά αυτή η παρατήρηση με την προστασία των δεδομένων, ε, πρέπει να πω ότι πρέπει λιγάκι να το δω το θέμα. Γιατί με την πρώτη ματιά, όσον αφορά τα θέματα της προστασίας των δεδομένων, δεν μου ήταν απόλυτα σαφής ο διαχωρισμός, αλλά εν πάση έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Νάταλη Γκρισμπέκ από την Άλντε. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και εγώ θα ήθελα ε, να επικροτήσω την επανέναρξη των συζητήσεων για αυτό το φάκελο, ε, για τον οποίο συζητήσει είχαν σταματήσει το 2013, όταν περιμέναμε ε, την ολοκλήρωση και την επίταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχει γίνει αυτό, ακόμα και αν έχει γίνει μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, μπορούμε τώρα να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την απαραίτητη μεταρρύθμιση. Γιατί θέλουμε την ε, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Eurojust. Ε, Ιδίω τώρα που η εγκληματική δραστηριότητα λαμβάνει όλα και πιο διασυνοριακές διαστάσεις και υπάρχει προσταθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Βος που δημοσίευσε και πρόσφατα την έκθεσή του με πολύ λεπτομερή εργασία και με την ευκαιρία των ε, θερινών διακοπών ε, ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε μικρές επισημάνσεις και αλλαγές. Τρία στοιχεία θα ήθελα να επισημάνω για το Σεπτέμβρη. Το σχόλιο για την ίδια την έκθεση είναι ότι πράγματι Έχουμε απαραίτητες διευκρινήσεις, όπως ε, υπογραμμίσετε και εσείς αγαπητέ συνάδελφε, για να ορίσουμε δηλαδή πολύ συγκεκριμένα τις ε, αρμοδιότητες της εισαγγελία και τους επιμέρους ε, θεσμούς και οργανισμούς για να υπάρχει η σωστή προσέγγιση στο σύστημα. Στο ίδιο μικρό θα ήθελα ε, να χαιρετήσω την ε, διευκρίνηση των αρμοδιοτήτων και της Eurojust και από την άλλη και της ε, εισαγγελία, γιατί δεν είναι τόσο απλό και πρέπει πολύ προσεκτικά να οριοθετήσουμε τις αρμοδιότητες αλλά και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις, αποφεύγοντας πάντα τις αλληλεπικαλύψεις. Μερικές παρατηρήσεις ακόμα, πολύ γρήγορα, που σίγουρα θα εντάξουμε σε τροπολογίες. Είναι αρκετά προβλέψιμο ότι η ομάδα μου θα δώσει μεγάλη έμφαση προκειμένου το σύστημα αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο ευρωπαϊκό και πιο κοινοτικό, για να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία. Μετά για τα ζητήματα δικονομίας και προσωπικών δεδομένων ε, σίγουρα θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στην Άλντε. Και τέλος, νομίζω ότι το, το θίξατε κι εσείς Άξελ, πώς ε, θα συνεργαστούμε με, και με τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην εισαγγελία και με τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στην εισαγγελία, προκειμένου όλα να κυλήσουν ομαλά και να υπάρχει ευρύτερη δυνατή προστασία παρά τις ε, διαφορές που αναδείξατε κι εσείς στις συμπεράσματά σας. Αυτά σε εδρές γραμμές θα θέλαμε εμείς ε, να εξετάσουμε ως πολιτική ομάδα. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά πυκνή αλλά και σαφέστατη αυτή η έκθεση. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ Ναταλή. Μουτζεντόφσκι παρακαλώ από το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Sprawozdawcy για πολύ e, e, wnikliwy ράπορτ. E, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Το θέμα είναι πολύπλοκο. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως όργανο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να ορίσουμε τις αρμοδιότητές της. Καταρχήν, αλλά Συγγνώμη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τις αρμοδιότητες του Eurojust πρώτα και όχι με την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να πούμε ότι είναι το, η παράνομη διακίνηση κλπ. Να ορίσουμε ποιες είναι οι αρμονότητε του Eurojust και μετά να περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεδομένου ότι ε, κάποια κράτη-μέλη δεν ε, έχουν συνυπογράψει τη δημιουργία τη ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Eurojust θα εξακολουθήσει να έχει πλήρες αρμοδιότητες. Είναι ένα ευρωπαϊκό όργανο που έχει πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη από, από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τις συνθήκες. Αντιλαμβάνουμε βέβαια ότι ο εισηγητής ε, κάνει εδώ ε, μια παρουσίαση και των δύο απόψεων. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, αναφορά στην οικοδόμηση, θεσμική, εσωτερική θεσμική οικοδόμηση της Eurojust. Μιλά για την ε, ευρωπαϊκή συνεργασία και στην εμπιστοσύνη ε, που πρέπει να δείχνουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να λειτουργεί σωστά η Eurojust. θα πρέπει να λάβουμε ε, επίσης υπόψη την άποψη των μελών που έχουν αυτοεξαιρεθεί, τη ε, Δανία και την Ιρλανδία δηλαδή. Ε, χώρες για τις οποίες χρειάζεται ιδιαίτερη σχέση προκειμένου να διαχειριστούμε τα θέματα αυτά καλύτερα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. για να Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εξ ονόματο και τη συναδέλφου Εύα Ζολή, με την οποία συνεργαζόμαστε πολύ στενά ε, για αυτό το φάκελο. Θα, θα ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, για το σχέδιο έκθεση. Η Eurojust όντω είναι απαραίτητο εργαλείο για να βελτιώσουμε την συνεργασία, τη δικαστική συνεργασία ε, μεταξύ των κρατών μελών. Συμφωνούμε ότι η αναθεώρηση τη Eurojust θα πρέπει να συνάδει και και να ευθυγραμμιστεί με την μελλοντική Ευρωπαϊκή Συγγελία προκειμένου να αποτρέψουμε ε, τυχόν καθυστερήσεις ό,τι αφορά την ε, θέσπιση αυτού του νέου οργανισμού. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ευθυγράμμιση και μεταξύ των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Eurojust, ακριβώς να προσδιορίσουμε πολύ συγκεκριμένα τον συντονισμό μεταξύ των δύο και να αποφύγουμε τυχόν συγκρούσει μεταξύ του. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων και μια ειδική σχέση, για παράδειγμα μέσω τη συνεργασία σε συναντήσει και ανταλλαγή ε, υποθέσεων και στοιχείων. Πρέπει λοιπόν από κοινού ε, να εργάζονται για να καταπολεμήσουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά ε, το οργανωμένο έγκλημα. Λυπούμαστε που έχουμε αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο για τους κανόνες Προστασία δεδομένων, όπως και για τους υπόλοιπους οργανισμούς και ελπίζουμε ότι κατά την εξέταση αυτού του φακέλου ήδη θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και στο νέο πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για προστασία δεδομένων. Από πλευρά μα, στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως ισχύει και για, τα, ε, και για τους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε αυτά να τα συνδυάσουμε εδώ σε αυτόν τον κανονισμό, αυτό που δεν καταφέραμε ε, στον κανονισμό Europol και Frontex μέχρι τώρα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, τις τροπολογίες μας και ε, προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα και ο Πρόεδρος. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Βόσου. No, I don't. I go to the commission. Α, όχι, συγγνώμη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσουμε το λόγο. Συγγνώμη, Άξελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή. πολύ δουλειά που έχει κάνει για την προετοιμασία αυτή της έκθεσης, το γνωρίζουμε καλά. Και με ασφάλεια μπορώ να πω ότι συμφωνούμε εν γέννη με τα όσα προτείνονται. Δεν μπορώ να σχολιάσω όλες τι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί προφανώ. δεν έχω αρκετό χρόνο. Δύο θέματα πολιτική φύσεως, δύο θέματα αρχή περισσότερο θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτον, Όταν προετοιμάσαμε την πρότασή μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εσωτερική δομή της ε, υπηρεσίας, ε, προφανώς βασιστήκαμε στην κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, τις οποίες συμφώνησαν τα τρία ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Αυτή η κοινή προσέγγιση είχε ως στόχο να εξασφαλίσει μια συνέπεια και μια συνέχεια στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται για όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ένα από τα βασικά σημεία αυτής της κοινή προσέγγισης είναι ότι η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στο υψηλότερο επίπεδο ε, λήψη αποφάσεων ε, σε κάθε μια αυτές τις υπηρεσίες. Ε, στην Eurojust αυτό είναι το συλλογικό όργανο και στα εκτελεστικά συμβούλια όπου αυτά υπάρχουν. Ο κ. Βος λέει ότι ε, η Κομισιόν βρίσκεται στο εκτελεστικό συμβούλιο και γι' αυτό λόγο δεν χρειάζεται να είναι ε, παρούσα στο συλλογικό όργανο. Όμω το εκτελεστικό συμβούλιο απλώ προετοιμάζει τι αποφάσει που θα λάβει το συλλογικό όργανο και η Κομισιόν θα πρέπει να είναι παρούσα και στο συλλογικό όργανο όπου λαμβάνονται αποφάσει. Αυτά σε ό,τι αφορά την ε, θεσμική πτυχή του ζητήματος, σημαντική και αυτή όμως και θα τεθεί στον τριμερή διάλογο στις Βρυξέλλες. Ένα άλλο θέμα αφορά την προστασία των δομένων Και εδώ συμφωνούμε με τον κύριο Άλμπρεχτ μάλλον. Ε, ε, επιθυμείτε να ακολουθήσουμε μια κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των δεδομένων για όλες τις υπηρεσίες. Και Πράγματι, όλα τα δεδομένα τα οποία εξετάζεται η Eurojust θα πρέπει να υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς προστασίας ε, με όλες τις υπόλοιπε υπηρεσίες και οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βέβαια, μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες συμπληρωματικές διατάξεις σε σχέση με αυτούς τους κανόνες και τις συμπεριλάβαμε ε, στις προτάσεις μας. Το θέμα συνδέεται ε, και με τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνονται για την συνέχεια που θα δοθεί στον κανονισμό 45 του 2001. Στον κανονισμό δηλαδή που θα αντικαταστήσει το 45 του Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βος λοιπόν. Θα συνεργαστούμε μαζί του και με τους υπόλοιπου συναδέλφου, ε, στο πλαίσιο του τριμέρους διαλόγου. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον ε, εισηγητή για την τελευταία του τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης και όλους τους συζητητές για αυτά που μας είπανε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε, δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω. Να πω μόνο ότι το όλο θέμα το αναβάλαμε μέχρι το Σεπτέμβριο και αυτό νομίζω ήταν ένα πολύ καλό βήμα για να μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα με την ησυχία μας. Και βεβαίως και χάρη της καλής δουλειάς της ε, γραμματείας ε, θα χάσουμε μόνο 10 μέρες σε όλη αυτή τη διαδικασία παρότι προστίθενται πολλές εβδομάδες. Δέκα μέρες όμως θα χάσουμε. Ευχαριστώ πολύ τη Γραμματεία για την πρόταση που κατέθεσε. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, νομίζω ότι ε, στην προστασία αυτή θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τα δεδομένα της Europol και της Eurojust. Εδώ ε, υπάρχουν ε, δύο ειδών δεδομένα, άρα δηλαδή θα πρέπει κανείς να δει ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Και αν τα μοιράσει κανείς με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ε, η Eurojust να ασχολείται με τα επιχειρησιακά δεδομένα, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο να καταθέσουμε μία σχετική πρόταση. Και αυτό έχει και νόημα από πλευράς ε, ουσίας, διότι η Eurojust ε, ε, ζει από την εμπιστοσύνη των κρατών μελών και της, των εισαγγελέων. Αλλά ίσως όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε και με περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως εγώ σας προειδοποιώ και λέω δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί ε, παρότι θα μπορούσε κανείς να νιώθει αυτό τον πειρασμό. Εγώ είμαι υπέρ της ε, διαφοροποίησης σε αυτόν τον τομέα έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες. Όσον αφορά το άλλο θέμα που έθιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να σας πω ότι έχω κάποια κατανόηση ότι και εκεί ε, θέλουν να τα κάνουν όλα ίδια. Μόνο που θέλω να πω ότι η κατάσταση στις ε, ε, υπηρεσίες ε, δίωξης ε, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες αυτές που επικρατούν οι συνθήκες όπως τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας και ακριβώς όπως είχαμε προβλέψει και για τη Europol να υπάρχει σχετική προσαρμογή. Κατά τα άλλα χαίρομαι για την μελλοντική συζήτηση το Σεπτέμβρη και χαίρομαι επίσης για το ότι τότε θα σκεφτούμε πώς θέλουμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν ε, όλοι μας ε, προσπαθούσαμε να αναζητήσουμε το συμβασμό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να στηριχθούν και έτσι και αλλιώ ε, θα ξανασυζητήσουμε στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σα και τη δική σα και των εισηγητών για αυτό το ζήτημα. Επιστρέφουμε στο χρονοδιάγραμμά μας τώρα. Περνάμε στο σημείο 6. Τα σημεία 6, 7 και 8 από κοινού. Α, 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για το θέμα της Eurojust. Περνάμε στα σημεία 6, 7 και 8. Τρία, ε, τρεις φάκελοι για το σύστημα πληροφοριών Schengen. Ε, θα κάνουν την παρουσίαση εισηγητές κ. Σκοέλιο και Λέιναρτς. Θα τους δώσω καταρχήν το λόγο ε, και μετά θα περάσουμε στην ε, Κομισιόν και τους εισηγητές ε, και τους χιώδεις. Ο κ. Κοέλιο καταρχήν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις στα πορτογαλικά. Το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν είναι η καλύτερη βάση δεδομένων ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει 70 εκατομμύρια alerts από ε, ε, σκάφη και χήματα που έχουν κλαπεί μέχρι, σώτου, μέχρι εξαφανισμένα άτομα υποστηρίζει τελωνιακές ε, και δικαστικές αρχές καθώς επίσης και την αστυνομία, συνοφυλακή ε, και ακτοφυλακή των κρατών μελών. Τέσσερα εκατομμύρια ε, αναζητήσεις έκαναν τέτοιου είδους αρχές στο σύστημα πληροφορίας Σέγγεν. Είναι κεντρικό κρίσιμο στην διατήρηση της ζώνης Σέγγεν. Το σύστημα καταμερίζει πληροφορίες και alerts ε, μεταξύ ε, αστυνομικών και δικαστικών αρχών, προστατεύει τα εξωτερικά μας ε, σύνορα και συνεισφέρει σημαντικά στην εσωτερική μας ασφάλεια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταρρυθμιστεί το σύστημα αυτό και να προσαρμοστεί στις σημερινές προκλήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις που έχει υποβάλει, αλλά είναι δυνατόν να, να βελτιωθούν. Αυτές τις προτάσεις ε, θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή. Το SIS μπορεί να συνεισφέρει στο να επιταχυνθεί και να είναι πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος. Ε, τα κράτη-μέλη για αυτό τον λόγο θα πρέπει να ε, εισάγουν στο σύστημα SIS ε, ε, ταχύτατα όλες τις προφορίες και να τις μοιράζονται με τη Europol. Αυτό θα προστατεύσει τα παιδιά μας, ήδη και ήδη τα προστατεύει, αλλά μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Ε, παιδιά που κυδεύουν να παχθούν, παιδιά τα οποία έχουν εξαφανιστεί, μετανάστες ή όχι, όλα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο SIS. Ε, το ότι κάποιο διασχίζει κάποια σύνορα δεν σημαίνει ότι μειώνεται η προστασία του. Είναι πολύ σημαντικό το σύστημα αυτό και για την ασφαλεία μα. Χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και έχει όλο και πιο σημαντικέ πληροφορίε. Θα πρέπει η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ε, να ε, είναι ικανή να δώσει απαντήσει και γι' αυτό όλο θα πρέπει να ενισχύσουμε το κεντρικό σύστημα και την προστασία του έναντι εξωτερικών επιθέσεων και αδυναμιών. Παραλλήλως, ε, θα πρέπει ε, να ε, προχωρήσουμε στην δημιουργία του SIS-2 με βελτίωση της προστασίας των δεδομένων και εξασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης, ε, χρηματοδότησης, επαρκούς χρηματοδότησης ενημέρωσης του κοινού. θα πρέπει από το ΣΥΣ1 στο ΣΥΣ2 να περάσουμε σταδιακά και προγραμματισμένα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και τις ελευθερίες. Επιστρέφω στα αγγλικά με τις προτάσεις μου. Ε, οι προτάσεις μου εστιάζουν σε τρεις άξονες. Ε, πρώτον, ε, όπως γνωρίζετε, το SIS είναι κεντρικό σύστημα. Έχει μία κεντρική βάση δεδομένων στο, στο και μία άλλη στην Αυστρία. Η Κομισιόν προτείνει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ένα εθνικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων που θα συνδέεται με το κεντρικό σύστημα. Εγώ αμφιβάλλω για το κατά πόσο αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Το Κοινοβούλιο πάντοτε εξέφρασε επιφυλάξεις για αυτή, για αυτή τη λύση. Και μέχρι τώρα η Κομισιόν δεν έχει καταφέρει να μας ε, δώσει μια εξήγηση για αυτήν την αλλαγή πολιτικής. Στο SIS 1 και το SIS 2 ακόμα και η Κομισιόν ήταν αρχικά ε, αντίθετη με αυτή την ιδέα. Επιπλέον αυτή η βρυδική λύση με κεντρικό επίπεδο και εθνικά επίπεδα δεν ακολουθείται σε κανένα άλλο μέσο όπως το ETS ή το Entry-Exit. Ούτε και φαίνεται να είναι συνεπές με τις ε, προτάσεις που απορρεούν από την ομάδα υψηλού επίπεδου για τις ανταλλαγές πληροφοριών. Προτείνω, όπως κάναμε και στο παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχτεί τον ισχύοντα συμβασμό. Τα κράτη-μέλη δηλαδή τα οποία θέλουν να έχουν ε, ένα εθνικό αντίγραφο να τους επιτρέπεται, αλλά αυτά τα οποία δεν το επιθυμούν να μην είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν ένα εθνικό αντίγραφο. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να εξασφαλίσουμε ότι το κεντρικό σύστημα θα μπορέσει να ε, υλοποιήσει όλα όσα του έχουν ανατεθεί. Γι' αυτό το λόγο ζητώ την ενίσχυσή του. Πώς? Αναπτύσσοντας μια ε, δραστήρια, μια λύση σύμφωνα με την οποία το σύστημα του Στρασβούργου θα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα της Αυστρίας. Έτσι θα ε, αυξήσουμε την ε, αποτελεσματικότητά του, την ταχύτητά του ε, και την ανθεκτικότητά του. Επίσης θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες σύνδεσης του κεντρικού συστήματος με τα εθνικά με τις εθνικές μονάδες. Ε, θα πρέπει να δώσουμε σημασία και σε αυτό έτσι ώστε η σύνδεση να είναι απρόσκοπτη. Προτείνω λοιπόν να, ε, να ε, διπλασιαστεί και η τηλεπικοινωνία και σύνδεση μεταξύ κέντρου και περιφερειών. Επίσης, το η Λίζα θα πρέπει να ενισχυθεί σύμφωνα με τη νέα του νομική βάση. Δεύτερον, ε, απάντηση στην τρομοκρατία. Η Κομισιόν εισάγει την υποχρέωση ε, να εισάγονται ειδοποιήσεις, alerts σε, οποιαδήποτε θέματα, σε οποιοδήποτε θέμα ε, έχει σχέση με την τρομοκρατία. Το πρόβλημα όμως είναι, έγκυται και στον τύπο και τον, τον όγκο των πληροφοριών που εισάγονται όταν δημιουργείται μια ειδοποίηση. Θα ήθελα να ζητήσουμε ε, να αναφέρεται στην ειδοποίηση και ο τύπος του αδικήματος. Και επίσης υπάρχει και ένας καινούριος τύπος ειδοποίησης, ε, ο, το, ο έλεγχος αναζήτησης, inquiry alert. Ε, αφορά ε, κάποιους συγκεκριμένους ελέγχους και παρόλο που είναι μία ε, το S IS αποτελείται από ένα σύνολο εθνικών βάσεων δεδομένων, στις οποίες δίνουμε πρόσβαση σε αλλοδαπούς σε, ξένα, σε άλλες χώρες. Οπότε, ε, πολύ συχνά κάποιες, κάποια κρατημέλη δεν μπορούν να φέρουν σε πέρα σε αυτό που τους ζητείτε. Οπότε, ε, ζητώ τα inquiry text, tests να είναι υποχρεωτικά. Ε, ο περιορισμό αυτών θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικέ περιστάσει και σε ειδικέ ε, επιχειρησιακές συνθήκες. Όπως σας είπα, το SIAS είναι εθνική βάση δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μοιράζονται όσε προφορίες χρειάζονται. Όμως πολλές συχνά χρειάζονται και προφορίες οι οποίε δεν βρίσκονται αποθηκευμένε στο σύστημα. Γι' αυτό το λόγο τα εθνικά ε, σημεία αναφορά. Ε, επικοινωνία, συγγνώμη, επαφή, θα πρέπει να δίνουν περισσότερε πληροφορίε, πρόσθετε πληροφορίε, όπω το απέδειξαν οι πρόσφατε τρομοκρατικέ επιθέσει που δημιούργησαν ανάγκη μεγαλύτερη πληροφόρηση, έκτακτη πληροφόρηση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι απαντήσει να γίνονται πιο γρήγορα, από 12 να μειωθεί το όριο σε 6 ώρε. και άμεση, και η απάντηση να είναι άμεση σε περιπτώσει τρομοκρατία. Ε, είναι πολύ σημαντικό το SIS στην καταπολέμηση τρομοκρατίας. Δίνει ποιοτικέ πληροφορίε στα κράτη-μέλη, αλλά μπορεί να ε, δώσει πληροφορίες και στις ε, μονάδες διάσωσης επιτόπου. Γι' αυτό το λόγο οι απαντήσεις θα πρέπει να δίδονται αμέσως κάθε φορά που μια εθνική αρχή μέσω του SIS εισάγει αναζητήσεις σχετικές με την τρομοκρατία. Όπως ζητήθηκε από τον κύριο Ντεπρέ σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Τρίτον, προστασία των παιδιών και μετανάστευση. Και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα παιδιά μας προστατεύονται. Γι' αυτό το λόγο προτείνω, αν ένα παιδί εξαφανιστεί, τα κράτη-μέλη να πρέπει ε, να εισάγουν ε, μία ειδοποίηση στο SIS. Επίσης να έχουμε ένα ειδικό τύπο ειδοποίηση που θα είναι αυτός που θα αφορά τα εξαφανισμένα παιδιά. Γιατί το 2015 μόνο, κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ευρωπόλ έλαβε 10.000 ειδοποίησει για εξαφανισμένα παιδιά. Οπότε προτείνω να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη ειδοποίηση για τα εξαφανισμένα παιδιά σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Eurodac να δημιουργηθεί μια τέτοια ειδοποίηση σε περίπτωση εξαφανισμένων παιδιών. Τέταρτον, υπηρεσίες. Να διασφαλίσουμε ότι και οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την βάση δεδομένων. Ε, η Europol βέβαια αλλά και η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Ακτιτοφυλακή. Η νέα Frontex ιδιαίτερος θα πρέπει να έχει πρόσβαση και στα hotspot. Πέμπτον, ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν της προτάσεις της φαίνεται να αγνοεί ότι το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη σε αυτά τα θέματα. Οποιαδήποτε θέματα δεν καλύπτονται από την πρόταση θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ε, εφαρμοστικών πράξεων στα οποία, στις οποίες το Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, χρήση βιομετρικών στοιχείων, αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους βιομετρικά στοιχεία όπως DNA κλπ, προτείνω ε, η χρήση τους να αποφασιστεί με, ε, μέσω της ε, ε διαδικασίας ε, των κατεξουδότησης πράξεων. Έκτον, αποτελεσματικότητα. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Το SIS ήδη βοηθάει την αστυνομία και τη συνοροφυλακή επιτόπου. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την επόμενη δεκαετία προκειμένου να εισαχθούν τα νέα ε, οι νέες διευκολύνσεις. Ε, η Κομισιόν αφήνει την προθεσμία ανοιχτή. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δεκτό. Ε, τα νέα χαρακτηριστικά του συστήματος θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί, να έχουν ενταχθεί 12 μήνες μετά την υιοθέτηση της πράξης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στη νομική βάση του SIS2 και να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου κατά τη στιγμή της υιοθέτησης του SIS2. Ε, το SIS είναι ε, ένα από τα, ε, λιγότερα, από τα συστήματα που λιγότερο έχουν αξιολογηθεί στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να αξιολογηθεί περισσότερο. θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει καινούριε προκλήσεις ε, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερα προστατωμένη αυτή παρουσίαση. Ο κύριος Λενάρτς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω για την πρόταση εισαγωγή ε, των ειδοποιήσεων για τις αποφάσεις επιστροφών στο σύστημα Schengen, SIS. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η βελτίωση του συστήματος ε, προκειμένου να υπάρχει και εμπιστοσύνη του κοινού σε ό,τι την πολιτική μετανάστευση στο σύνολό τη. Γιατί αν θέλουμε ή μάλλον τώρα που αποτυγχάνουμε στις ε, επιστροφές το 60% τελικά οι πραγματικοί πρόσφυγες, αυτοί που προσπαθούν να ξεφύγουν από την ε, από τον πόλεμο ε, θα είναι αυτοί που θα πληγούν τελικά γιατί δεν θα έχουμε τη, τα μέσα ε, να τους προστατεύσουμε όπως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό. Χαιρετίζω λοιπόν την ε, πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή αυτών των alerts για να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Είναι ένα μικρό αλλά κρίσιμη σημασία βήμα. Και υπάρχουν και ορισμένε παρατηρήσει που έκανα και στο σχέδιο έκθεση. Πρώτον, επικαιροποίηση τη πρόταση τη Επιτροπή για τα πρόσφατα ε, υιοθετημένα κείμενα όπως είναι ε, η ανακοίνωση για τρομοκρατία σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση μιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Η Κομισιόν δίνει μεγάλο ε, πεδίο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να ορίσουν μια αρχή και καθώς ήδη στο Σέγγεν υπάρχει ένας κατάλογος ε, αρχών που συνεργάζονται πολύ καλά, καλύτερο θα ήταν εκεί να γίνεται, με αυτές δηλαδή τις αρχές να γίνεται ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών για τις αποφάσεις επιστροφών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην προσθέσουμε ε, ε γραφειοκρατικό άχθος, όλη αυτή η διαδικασία να παραμείνει αποτελεσματική. Οπότε, για τα άτομα που ε, συλλαμβάνονται στα σύνορα και δεν εισέρχονται δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν χρειάζεται να μπουν τα δεδομένα αυτών των ατόμων στο Σέγγεν. Το ίδιο όταν οι αρχές εντοπίζουν άτομο που δεν έχει ακολουθήσει την προθεσμία για να αποχωρήσει, αλλά ακολουθεί κάνει κάτι διαδικασία τότε δεν χρειάζεται και πάλι να μπει στο σύστημα SIS. Μία απλή επιστροφή, μάλλον επιβεβαίωση της επιστροφής αρκεί. Και κάτι ακόμα για την αποτελεσματικότητα. Το σύστημα SIS είναι ένα σύστημα που βασίζεται στις ενέργειες. Όταν τα κράτος μέλος αποφασίζει να αναστείλει ε, μία απόφαση επιστροφής, καλό θα ήταν και το alert να είναι προσωρινά διαθέσιμο για να μην ε, μπερδεύει αυτό τις άλλες αρχές που μπορεί να εντοπίσουν αυτό το πρόσωπο. Κάτι άλλο πιο περίπλοκο ενδεχομένω και πάλι για το Κοινοβούλιο είναι το θέμα της διατήρησης των δεδομένων. Στην μελέτη σκοπιμότητα που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρχε επιλογή ε, να διατηρούνται τα ε, δεδομένα για μια περίοδο πέντε ετών. Στην πρόταση η Επιτροπή αποφάσισε να μην κάνει κάτι τέτοιο, αλλά να διαγράφονται απευθείας όλα τα δεδομένα όταν φύγουν αυτά τα άτομα από την επικράτειά μας. Εγώ διαφωνώ με αυτή την επιλογή. Έχω επανεισάγει την ε, πενταετή αυτή περίοδο. Θεωρώ ότι είναι σημαντική ε, για να παραμείνει χρήσιμο το σύστημα. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα για την πρόταση της Κομισιόν. Κάτι το οποίο παρατήρησα στις συζητήσεις μου ε, σχετικά με, τις, ε, με το σύστημα SIS και τις αποφάσεις περί επιστροφών. Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια ε, πιο υπόγεια προβλήματα σε διαφορά τη συνεργασία στον τομέα των επιστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό εξίσου να εξετάσουμε και πάλι την ίδια την οδηγία επιστροφών και να σιγουρευτούμε ότι κάποια από τα ε, ζητήματα αυτά που δυσχεραίνουν τη συνεργασία να τα εξετάσουμε σε μία αναθεωρημένη πρόταση περί της οδηγίας επιστροφών. Αυτό λοιπόν καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στους κοιόδης, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία. Παρακαλώ, κυρία Τζάνσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο και τον κύριο Λέναρτς για την ε, πολύ ε, θετική και επικοδομητική πρόταση. Νομίζω ότι θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις. Δεν ε, μπορώ να βρω κάποιο σημείο στον οποίο να διαφωνούμε. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή βάση συζητήσεων. για αυτό το μελλοντικό διάλογο. Συμφωνώ κύριε Κοέλιο με τις παρατηρήσεις σας. Μάλιστα εσείς ε, ενισχύετε από πολλές απόψεις την πρότασή μας. Ήμασταν πιο επιφυλακτικοί γιατί ξέρουμε τα όρια των κρατών μελών. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή προφορίων με την Europol ή για αυτόν τον περιορισμό των 12 ωρών ε, στην απάντηση, ξέρουμε, για παράδειγμα, και τις 12 ε, ώρες, γιατί η απάντηση ε, προκύπτει κατόπιν διαβούλευση και με πολλές διαφορετικές υπηρεσίες ε, και αρχές. Γι' αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν ε, εντός 12 ώρων ή και λιγότερο. Όμως ξέρουμε ότι σε ζητήματα που άπτονται της τρομοκρατίας, εκεί η απάντηση πραγματικά είναι άμεση και παίρνουν πολύ στο σοβαρά αυτές τις περιπτώσεις. Όπως και να έχει εμείς βεβαίω θα το συζητήσουμε λεπτομερώς και με συγκεκριμένα παραδείγματα προκειμένου να ενισχυθεί και η ικανότητα αυτών των αρχών ε, για να ανταποκρίνονται το στομότερο δυνατόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων και τα θέματα μετανάστευσης, και εδώ συμφωνούμε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικες, ανήλικοι συγγνώμη, θα πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερως και να γίνονται ορατοί στο σύστημα, εδώ προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και το θέμα της, ε, των αόρατων ανηλίκων, που είναι γι' αυτό σημαντικό πρόβλημα. Ένα από τα πράγματα που θα μας βοηθήσουν θα είναι τα δεκτυλικά αποτυπώματα. Εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε πραγματικά ε, με τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ε, τα δεκτυλικά αποτυπώματα αυτών των ανηλίκων. Ιδάλλως δεν θα μπορούν να εντοπιστούν, να ταυτοποιηθούν εάν παρουσιαστούν με διαφορετικό όνομα. Και θα ήθελα να θίξω κάτι ακόμα που αναφέρατε και εσείς στο θέμα των εθνικών αντιγράφων έναντι του πλήρως ε, ε, κεντρικού συστήματος. Θα ήθελα να πω ότι το SIS είναι η μοναδική βάση δεδομένων ασφαλεία στην Ευρώπη. Δεν είναι βάση δεδομένων μετανάστευση. Οι υπόλοιπε κεντρικέ βάσει δεδομένων στην Ευρώπη είναι όλε μεταναστευτικέ βάσει δεδομένων. Και η Eurodoc και το σύστημα εισόδου-εξόδου. Το ΣΥΣ είναι βάση δεδομένων ασφαλεία. Εάν δεν δουλέψει αυτή η βάση δεδομένων, μπορεί να χάσουμε ζωές ε, ή ζωέ η βάση δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα. Τότε ακόμα και συνοριακοί έλεγχοι μπορεί να επανεισαχθούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα του ΣΥΣ. Γι' αυτό και θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε και σε τεχνικό επίπεδο τη διαθεσιμότητα του ΣΥΣ. Λυπάμαι που καθυστερήσαμε να σας απαντήσουμε. Τώρα όμως ε, βρίσκεται καθοδόν αυτή η απάντηση που σας δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για το κατά πόσο το σύστημα δεν είναι διαθέσιμο σε κεντρικό επίπεδο. Όμω είναι μια πολύ καλή βάση η συζήτηση σε αυτή, πώ μπορούμε δηλαδή να ενισχύσουμε το κεντρικό σύστημα και να δώσουμε και εναλλακτικέ λύσει στα κρατημέλη που δεν έχουν εθνικό αντίγραφο. Θα ήθελα όμω και πάλι να υπογραμμίσω ότι το σύστημα SIS χρησιμοποιείται σε διαφορετικές ε, συνθήκες και σε αυτό έχουν πρόσβαση διαφορετικές αρχές και είναι και τεχνικά περίπλοκο, οπότε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν εθνικό αντίγραφο ε, αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς στη χρήση του συστήματος, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα, για παράδειγμα, ε, να έχουν πρόσβαση στην αυτόματη αναγνώριση ε, πινακίδων, για παράδειγμα, ενός οχήματος. Αν δεν έχουν εθνικό αντίγραφο, λοιπόν, δεν θα τα βλέπουν όλα αυτά και μπορούν να αξιοποιήσουν τεχνικά πραγματικά αντίγραφα του συστήματος, γιατί έτσι κάνουν διάφορους ελέγχους και τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτών των τεχνικών αντιγράφων. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω και στον κύριο Λέναρτς για τις επιστροφές. Να τον ευχαριστήσω επίσης. Ήταν ε, ε σκόπιμη αυτή η απόφαση που ε, δεν προσδιορίσαμε μία ενιαία αρχή γιατί υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου δεν έχει την ε, πλήρη ε, αρμοδιότητα μόνο η αστυνομία για τις αιτήσει ασύλου και δεν, έχουν, δεν είναι λοιπόν αρμόδιες να τις διαχειριστούν. Και υπάρχουν και χώρες όπου η αστυνομία δεν έχει καν πρόσβαση στα στοιχεία μετανάστευσης και στις, στα συστήματα που διαχειρίζονται τις, τις επιστροφές. Γι' αυτό θα ήταν δύσκολο να έχουμε αυτή την τεχνική, τεχνικό σημείο επαφής με τις βάσεις δεδομένων μετανάστευσης. Γι' αυτό αφήσαμε ανοιχτή αυτή τη δυνατότητα κάτι μέλη να ορίσουν κάποια άλλη αρχή ασύλου, μετανάστευσης για να είναι το ενιαίο σημείο επαφής για τις υποθέσεις επιστροφών. Γιατί αυτοί έχουν τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Μιλήσατε κύριε Λέναρτς ε, για το σύστημα SIS που βασίζεται στις ενέργειες και συμφωνώ. Όμως υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Λέτε ότι για, τις, ε, για τα alerts ε, επιστροφών θα πρέπει να έχουμε το, την πενταετή διατήρηση των δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση για τους αξιωματούχους, αξιωματικούς στον δρόμο, αν το άτομο τίθεται το ζήτημα κατά πόσο έχει επιστρέψει νομίμως το άτομο, η πρώτη αντίδραση του αστυνομικού θα είναι ότι το άτομο αυτό παρανόμως βρίσκεται στην επικράτεια της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο να χρησιμοποιήσουμε άλλες βάσεις δεδομένων για να καταχωρήσουμε το ιστορικό ε, των ε, ατόμων που επιστρέφουν, όπως το Eurodac. Γιατί πρέπει και οι ίδιοι αξιωματικοί να ξέρουν ε, τι ε, άγουσαν να επιλέξουν για ένα άτομο. Και αν ε, παραμείνει μια ειδοποίηση επιστροφής στο σύστημα, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η επιστροφή Οπότε μπορεί τελικά ε, να θίγεται και το ίδιο το πρόσωπο, το οποίο να έχει επιστρέψει νομίμως στην επικράτεια, αλλά έχει, μετά χάνει αυτά τα δικαιώματα. Τέλος πάντων, ε, θα παρακολουθούμε προσοχή τη συνέχεια της συζήτησης και προβλέπουμε τη συνέχεια της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ. η Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο για την εξαιρετική γνώση του συστήματος SIS και επίσης και για τη δουλειά που έκαναν καταθέτοντας ε, τις προτάσεις. Όπως είπε και ο υπουργό μου κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό αντιμετωπίζει το σύστημα SIS ως μια προτεραιότητα και προχωράτε με ταχύτητα σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εκ μέρους της Προεδρίας εμείς θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις προτάσεις αυτές ως προτεραιότητα και δεσμευόμαστε πλήρως ε, να προχωρήσουμε το στεμό των ενετών με τις προτάσεις για το σύστημα SIS. Πιστεύουμε ότι ένα λειτουργικό SIS ε, βρίσκεται στην καρδιά της συνεργασίας του Schengen και παίζει σημαντικό ρόλο στο να διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Αυτό είναι μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος μας είναι μέχρι τον Οκτώβριο να έχει επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο, μετά στο Κοινοβούλιο και να αρχίσουν οι ε, διοργανικές ε, συζητήσεις το φθινόπωρο ίσως και να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του έτους να σας ενημερώσω λιγάκι για το πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Κατορτώσαμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο γύρο των συζητήσεων στο Συμβούλιο ε, στις αρχές Ιουλίου. Εξακολουθούμε να έχουμε ε, μέχρι τα τέλη Ιουλίου και άλλες ε, συναντήσεις για να πλησιάσουμε περισσότερο στην γενική προσέγγιση του Συμβουλίου. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο, παρότι βέβαια υπάρχει ακόμα δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαι αισιόδοξο ότι αν τελικά οι θεσμοί ε, οργανιστούν, εργαστούν σκληρά επί του θέματο, τότε μπορούμε και να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η συνεργασία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και αυτό ε, θα προσφέρει στους πολίτες αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Χαίρομαι που είστε αισιόδοξο, αλλά αν δεν είναι και κανείς αισιόδοξο όταν ξεκινά μια προεδρία, ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πάμε τώρα στους ε, σκιώτης από τους σοσιαλδημοκράτες πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ ε, τους δύο εισηγητές που παρουσίαν σήμερα την έκθεσή του. Εγώ ε, θα ξεκινήσω καταρχήν με το φάκελο που αφορά στη δουλειά του κυρίου Κοέλο. Το σύστημα Schenken, SIS, είναι από τα μεγαλύτερα συστήματα υπολογιστών στον κόσμο και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό για την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να διευκολύνεται η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων σε χώρο Σέγγεν. Χαιρετίζω γενικά την έκθεση του κυρίου Κοέλο που στόχος ε, είναι πιο αποτελεσματικό σύστημα αντικαθιστώντας ε, την σχέση, ε, αντικαθιστώντας όλα με μία άμεση διασύνδεση. Και επειδή το σύστημα SAS είναι ακρογωνιαίος λίθος για την ελεύθερη μετακίνηση, είναι επιτακτικό. Αυτό το σύστημα να είναι προσπελάσιμο ανα πάσα ώρα και στιγμή. Γι' αυτό και εγώ στηρίζω αυτά που είπατε, να ε, ενισχυθεί η υποδομή και το σύστημα να αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Βέβαια θέλω κάτι να πω, ότι όλα αυτά σημαίνουν οικονομική επένδυση και εδώ συμφωνώ ότι ένα μεγάλο σύστημα απαιτεί και μεγαλύτερη επένδυση. Αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό εγώ ε, θέλω να κρατήσετε ανοιχτή την επικοινωνία έτσι ώστε και όλοι μας να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση που θα τη δεχτούν όλοι. Να πω και κάτι σχετικά ε, με κάτι που υπογραμμίσατε ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν θέλουν, που δεν θα θέλουν εθνικό αντίγραφο, ε, δεν θα πρέπει και να το ε, κατασκευάζουν να είμαστε όλοι στην ίδια άποψη, της ίδιας άποψης όσον αφορά αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό. Και κάτι άλλο. Καταρχήν στηρίζω αυτό που ζητήσατε να υπάρχουν ιδιώτες μηχανικοί οι οποίοι ε, θα διασφαλίζουν τα συστήματα και επίσης και το ποιος θα έχει πρόσβαση στα συστήματα. Βεβαίω να επισημάνω ότι η δική μου πολιτική ομάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε αυτό να συμβαδίζει με το πακέτο προστασία δεδομένων που εγκρίθηκε πέρυσι και κάτι άλλο. Έχουμε ανησυχίες σχετικά με το να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη εξωτερικούς ανάδοχους. Αλλά Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα στηρίξουμε τη δική σας την προσέγγιση. Και οφείλω επίσης να υπογραμμίσω ότι εμείς ως ασχελοδημοκράτες εξακολουθούμε να ανησυχούμε σχετικά με τη χρήση βιομητρικών δεδομένων του DNA και των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ε, και στηρίζουμε ε, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτές οι καταχωρήσεις για αγνοούμενους ε, αυτές οι ανακοινώσεις θα πρέπει να βασίζονται σε πολύ ξεκάθαρα κριτήρια. Ε, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να μας δώσει κάποιες περισσότερες προφορίες ε, για το θέμα των ανακρίσεων. Αυτό θα μας έδινε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης και έτσι θα μπορούσαμε και εμείς να τοποθετηθούμε πολιτικά επί του θέματος με μεγαλύτερη διαφάνεια. Και δύο άλλα θέματα που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Ο εισηγητής σε κάποιο σημείο προτείνει κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το εγχειρίδιο. Αυτό το στηρίζουμε και είναι πολύ σημαντικό και το ότι ε, θέλετε να καταθέσετε ε, τροπολογίες για την εκπαίδευση υπαλλήλων που χρησιμοποιούν το σύστημα SIS. Ε, τώρα, όσον αφορά την άλλη έκθεση, για μας είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε αποφάσεις για επιστροφή να μην εμφανίζονται, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα επιβαρύνει το σύστημα με τις ανακοινώσεις για αγνοούμενους που είναι ήδη επιβαρημένο. Θα καταστήσουμε, θα καταθέσουμε ε, προτάσεις για το θέμα αυτό. Και ξέρουμε και ότι ε, ο εισηγητής προτιμάει τα δακτυλικά αποτυπώματα για υπηκόους τρίτων χωρών. Ίσως μπορεί ο εισηγητής να μας εξηγήσει λιγάκι καλύτερα τη θέση του για την προτινόμενη τροπολογία ε, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Το στηρίζουμε γιατί μοιάζει να είναι θετική εξέλιξη, κυρίως όσον αφορά του υπηκόους τρίτων χωρών, όταν ε, ε, γίνεται κοινή χρήση των πληροφοριών για τα άτομα αυτά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι έτσι κάτι γενικότερο, πολιτικά γενικότερο. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου τα κράτη-μέλη καλούνται να αντιδράσουν μετά από αιτήματα άλλων τρίτων άλλων κρατών, αλλά το θέμα είναι ε, πότε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα έχουν την ίδια άποψη ε, έτσι ώστε κάτι που λέγεται να αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρετε, αυτό είναι ένα ερώτημα ε, που προκύπτει αν διαβάσει κανείς ε, την έκθεση Κομισιόν. Ευχαριστούμε τους ηγητές και προσβλέπουμε στη συνεργασία. Ο κύριος Ζεράρ Ντεπρέ από τους Φιλελεύθερους. Ε, Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι υπήρχε και άλλη μια ομάδα στον κατάλογο πριν από μένα. Θα ξεκινήσω από την έκθεση Κοέλιο, τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Ε, στηρίζουμε τις γενικές ε, κατευθύνσεις της ε, πρότασης Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της λειτουργίας του SIS. Όμως, θα, υποβάλουμε και, θα υποστηρίξουμε και πάρα πολλές επιστροπολογίες του εισηγητή. Καταρχήν και εμείς έχουμε δισταγμούς σε ό,τι αφορά την υποχρέωση τα κράτη-μέλη να έχουν ένα εθνικό αντίγραφο. Προτιμούμε την αλλακτική της ενίσχυσης της υποδομής του κεντρικού συστήματος. Δεύτερον, στηρίζουμε τις τροπολογίες του εισηγητή που αφορούν την βελτίωση της πρότασης Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Τρίτον, και την, πρόσβασή του. Τρίτον, υποστηρίζουμε την πρόταση του εισηγητή έτσι ώστε το καινούριο SIS να ε, ξεκινήσει τη λειτουργία το συντομότερο δυνατό. Τέταρτον, στηρίζουμε το σύνολο των τροπολογιών του εισηγητή ε, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η πρόταση για τις ε, καινούριες απαιτήσει του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το, το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Πέμπτον, στηρίζουμε την τροπολογία του που αφορά την ε, τον αποκλεισμό της δυνατότητας στα κράτη-μέλη να μην κάνουν ελέγχους ε, έρευνας και αυτές να αντικατασταθούν από διακριτικούς ελέγχους γιατί η εθνική τους νομοθεσία δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί. Έκτον, Στηρίζουμε επίση την πρόταση του εισηγητή που προβλέπει στην περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών που σχετίζονται με την τρομοκρατία ε, η προθεσμία απάντηση να είναι μηδενική, δηλαδή να, γίνεται, να δίνεται άμεση απάντηση και όχι να δίνεται προθεσμία 12 ε, ωρών, διότι αυτή μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειε αυτή η καθυστέρηση. Ορισμένε παρατηρήσει. Πρόσθετε ε, συμμεριζόμαστε την ιδέα του εισηγητή να εναρμονίσουμε ακόμα περισσότερο την ε, εισαγωγή ε, μιας ειδικής καταχώρησης ε, για ατόμα τα οποία έχουν καταδικαστεί ε, σε ποινές φυλάκισης για σοβαρά δικήματα. Ως τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό. Όταν όμως προτείνει μια άρνηση εισόδου για μια καταδίκη φυλάκιση ενός έτους, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί γιατί οι ορισμένε χώρε είναι πολύ λίγο. Τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά τον κύριο Κόελιο. Ε, συμφωνούμε με την πρόταση να εισάγουμε καταχωρήσει για ε, μη συνοδευόμενου ανήλικου που έχουν εξαφανιστεί. Μιλώ για μετανάστε βέβαια. Ε, δεν ξέρω αν χρειάζεται μια ιδιαίτερη κατηγορία ε, καταχώρησης όταν πρόκειται για ανηλικούς, αλλά έχουμε και τις γυναίκες τις, οι, οποίες, ε, οι οποίες κινδυνεύουν αν επιστραφούν να υποστούν υποχρεωτικούς, υποχρεωτικούς ε, γάμους ή ακροτηριασμού γυναικείων οργάνων, γεννητικών οργάνων. Συγγνώμη. Ε, ενδεχομένως θα μπορούσαμε και τα δύο αυτές κατηγορίες να τις εντάξουμε στο ίδιο, στο, στην ίδια καταχώρηση alert. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση Λέναρτς, ε, πολύ καλή, αλλά και εδώ έχω ορισμένες παρατηρήσεις. Συμφωνώ με εκείνους που ε, εξέφρασαν επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τον, την υποχρεωτική διατήρηση πληροφοριών επιστροφών για πέντε χρόνια στο SIS. Για δύο λόγους. Πρώτον, όταν κάποιος έχει εκτελέσει την επιστροφή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει παραβεί τον νόμο. Ε, δεύτερον, οι σχετικές πληροφορίες για την εγκατάλειψη της επικράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται για πέντε χρόνια στο Eurodac. Αυτό το αποφασίσαμε τελευταία. Επιπλέον, σύντομα θα έχουμε και το σύστημα αιτίας. Δηλαδή, ε, προηγούμενη άδεια εισαγωγή, ε, εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συνδέεται με το Eurodac. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει επιστραφεί έτσι, θα έχει καταγραφεί στο Eurodac και δεν θα μπορεί να ξαναμπεί εύκολα αν δεν, αν δεν ε, το Eurodac. Ο εισηγητής προτείνει επίσης κάποιος ο οποίος κρατείται μέχρι τη μετακίνησή του να μην πρέπει να καταχωρείται στο SIS. Πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ιδέα. Ο εισηγητής προτείνει επίσης να μην επιτρέπουμε την εισαγωγή παρά μόνο των ε, δακτυλικών ε, ε, αποτυπωμάτων αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα, διότι θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατές ε, υπάρχουσες τεχνολογίες και να βελτιώσουμε τη διαλειτουργικότητα. Επίσης στηρίζω τις προτροπολογίες του εισηγητή, που έχουν ως στόχο να βελτιωθούν οι εγγύησεις ό,τι αφορά την ανταλλαγή πρόσθετων πληροφοριών με τρίτες χώρες. Όπως κάναμε και στο Eurodac. Ο εισηγητής προτείνει να γίνει υποχρεωτική παρουσία ε, ε δακτυλικού αποτυπώματος ή φωτογραφίας προσώπου όταν εισάγεται μια ε, καταχώρηση. Συμφωνώ απολύτως με αυτή την πρόταση. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Αυτές είναι οι απόψεις της ομάδας μου. Um, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους ε, σκιώδεις ε, για τις ε, λεπτομέρειες και τώρα θα ήθελα να επανέλθω στον κύριο Κοέλο να μας πει αν θέλει να κάνει κάποια τελικά σχόλια. Οι άλλοι σκιώδεις δεν ήταν παρόντες. Ε, πολύ σύντομα σχετικά με ορισμένα θέματα που εφήγησαν, λέει ο κύριο Λένερς, ε, το γιατί προτιμάμε τα δακτυλικά αποτυπώματα από την εικόνα, από τη φωτογραφία, είναι γιατί στην πρόταση δεν προβλέπεται καμία υποχρέωση ε, να μπείτε το ένα για το άλλο σε αυτές τις καταχωρήσεις εξαφανιστέντων, μάλλον αγνοωμένων. άρα δηλαδή είτε δακτυλικά αποτυπώματα, είτε φωτογραφίες, το προτιμούμε από το να μην είναι δεσμευτικά είτε το ένα είτε το άλλο. Εμείς προτιμούμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και όσον αφορά στο ε, ποια είναι η τελική απόφαση επιστροφής, ε, πώς μπορεί να γίνει αυτό λειτουργικό. Ξέρετε, ε, μπορεί ε, μία απόφαση να παραμείνει. Δεν μπορεί να φεσιβάλει όλες τις ε, αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στην ε, υποχρετική περίοδο κράτηση δεδομένων πέντε έτη, Γεράρ, ξέρεις, ε, αυτά τα δεδομένα θα υπάρχουν και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δίδονται θα είναι μέσα σε μία τράπεζα δεδομένων ε, και να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ε, τα δεδομένα αυτά. Ε, και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις και τις προτάσεις τους. Θέλω να σας πω ότι είχαμε ήδη τρεις συναντήσεις και οδών εισηγητών. Ε, προσβλέπω στη συνεργασία με όλους. Ε, σε αυτές τις ε, συναντήσεις ήταν παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστώ την Επιτροπή, κυρίως τη Σουζάνα, για τη συνεργασία που είχαμε για τη βοήθειά της. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα για όλους μας και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι το σύστημα SIS είναι καθοριστική σημασία για να προσφέρουμε ασφάλεια στους πολίτες μας. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Και νομίζω ότι με τη συνεισφορά όλων θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε, ο και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε τους οδηγητές, ε, την Επιτροπή, τους Σκεώδης ε, για τη δουλειά τους. Λοιπόν, συνάδελφοι, σήμερα το απόγευμα έχουμε πολλή δουλειά. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 9 που είναι μία παρουσίαση της Επιτροπής και αφορά στην εντολή της ε, για τη Frontex. Νομίζω ότι όλοι μας ε, θέλουμε αυτή η ε, Επιτροπή να λειτουργεί και πρόκειται για την τρίτη έξι επιτροπή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έδειξη λειτουργία τη φυλακή, ακτοφυλακή και όποιο θέλει μετά μπορεί να παρέμβει. Πρώτα η επιτροπή, νομίζω ο Σάιμον θα λάβει το λόγο. Okay, colleagues, if we're ready for the uh, presentation from the Commission on the operalization of the border guard, Simon, please. Good afternoon. Um, Καλησπέρα. Ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση για την πρόοδο που σημειώνεται σε ό,τι αφορά την θέσπιση της Ευρωπαϊκής ε, Συνοριοφυλακής και Εκτοφυλακής. Έχουμε την τρίτη και τέταρτη έκθεση όπου περιγράφουμε την κατάσταση και το Μάιο και τον Ιούνιο. Τα έχετε ακούσει δηλαδή αυτά. Θα είμαι λοιπόν σύντομος. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω εν συντομία τι έχει γίνει από τις αρχές Μαρτίου του 2017. Όταν ε, είχαν προετοιμαστεί οι προηγούμενες εκθέσεις. Θα ήθελα αρχικά ε, πραγματικά να ευχαριστήσω και να δώσω χαρητήρια ε, στους υπαλλήλους ε, της υπηρεσίας, γιατί πραγματικά έκαναν τη Frontex σε μια πραγματική, ε, ένα πραγματικό οργανισμό ακτοφυλακής, συνοριοφυλακής και είναι κάτι πολύ πρόσφατο. Ξεκαθαρίζω βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια και από τις δύο εκθέσεις γενικά προκύπτει ότι παρότι βλέπουμε μια συνεχόμενη βελτίωση και ανάπτυξη των ε, δραστηριοτήτων οργανισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου θεωρούμε ότι απαιτούνται βελτιώσεις και ε, καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών, ιδίω από τα κρατη και κάποιοι τομείς που χρήζουν ιδιαίτερης πολιτικής έμφασης. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή παρέχει επιχειρησιακή στήριξη επιτόπου στα κρατη σε ό,τι αφορά την διαχείριση σύνορων και αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1.600 συνοριοφύλακες και λοιπό προσωπικό που έχει αναπτυχθεί στην επικράτεια των κρατών μελών σε διάφορα τμήματα των εξωτερικών συνόρων. Και αυτό είναι προφανώς εντυπωσιακό, όμως ακόμα παραμένουν ορισμένα κενά που ε, εγείρουν ορισμένες ανησυχίες και εκεί θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ανάληψη δράσης από τα κράτη-μέλη. Τώρα, για λόγους ε, συντομίας, έχουμε κάποιους ε, τομείς προτεραιότητας, όπως είχαν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, δεν έχουμε πλήρη ικανότητα των ε, Rapid Reaction Pools. Εδώ υπάρχουν ε, λοιπόν περιθώρια βελτίωσης. Δεν είχαμε ε, τη συμβολή όλων των κρατών μελών, μόνο 14. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για τον εξοπλισμό ας πούμε, που δεν έχουμε, δεν έχουμε υπεράκτια σκάφη που να κάνουν περιπολίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά, αυτές τις ομάδες Rapid Reaction Pool, είναι ένα πρόβλημα, γιατί όταν ε, το είχαμε αποφασίσει, είχε ξεκαθαριστεί ότι θέλαμε 1.500 ε, συνοριοφύλακες κατονομασμένους όμως, που σε οποιαδήποτε κρίση να μπορούν να αναπτυχθούν. Μόνο εννέα κρατημέλη έχουν δώσει τα ονόματα αυτών των συνοριοφυλακών, από τις υπόλοιπες έχουμε λάβει υποσχέσεις, αλλά ε, από πλευράς χρονοδιαγράμματος είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια γενικόλογη υπόσχεση, παρά ε, να έχεις ε, κάτι, τα συγκεκριμένα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Οπότε ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό δεν το είχαν σε καμία περίπτωση στους νομοθέτες κατά νου όταν ε, συμφωνήθηκε. Ε, καταλήξαμε λέει, στη συμφωνία, και θα, το, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε επίπεδο υπουργών για τα συγκεκριμένα ονόματα αυτών των συνοριοφυλάκων, γιατί έτσι θα φροντίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν και την κατάλληλη κατάρτιση. Ο οργανισμός ε, έχει κάνει σημαντική δουλειά σε ό,τι αφορά την ε, πρώτη ε, αξιολόγηση των ευάλωτων σημείων κάθε κράτους μέλους. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν ε, και προκύπτουν οι συστάσεις. Προς το παρόν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που προτείνονται προς 20 κράτη-μέλη ε, για να καλύψουν αυτά τα ευάλωτα σημεία τους. Μετά, το επόμενο βήμα είναι πώς από την θεωρία να περάσουμε σε πραγματικές ε, ασκήσεις προσωμείωσης. Σε έξι κρατημέρια θα γίνει αυτό στο πρώτο στάδιο και έτσι θα είμαστε πολύ πιο ικανοί και προετοιμασμένοι στην αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων. Λέμε επίση ότι σε κάποιους ε, τομείς υπάρχει ενισχυμένη εντολή και αυτό του δίνει τη δυνατότητα ε, να κάνουν πολύ περισσότερα για να στηρίξουν ε, τα κρατη Και εσείς, ε, Πρόεδρε, παρευρεθήκατε στο άτυπο Συμβούλιο και, για παράδειγμα, για τις επιστροφές όταν συζητήθηκε το θέμα των επιστροφών, ο διευθυντής του οργανισμού είπε ότι ο οργανισμός πλέον μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στον τομέα των επιστροφών. Ήδη έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, αυξάνεται ο ρυθμός των επιστροφών αυξάνεται ο αριθμό και των ατόμων που περνούν από τη διαδικασία της επιστροφής, όμως ε, ακόμα πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν. Για σας εξίσου σημαντικό είναι η αναθεώρηση της στρατηγικής θεμελιωδών δικαιωμάτων του οργανισμού. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, υπάρχουν διαβουλεύσεις και με το Φόρουμ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, που μας έχει δώσει ορισμένες συστάσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους και την ε, αναγκαιότητα ειδική ε, εστίασης σε ζητήματα προστασίας ε, ανηλίκων. Κάτι άλλο είναι ο μηχανισμός ενστάσεων Εκείνο είναι αυτό κάτι το οποίο μας προβληματίζει στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, για... προτείνω να είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί το επόμενο θέμα είναι οι ε, συζητήσεις με τη Σερβία. Να σας πω μόνο ότι έχουμε εντολή διαπραγματεύσεων και με την πρώην Ιγκοσλοβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όμως δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις λόγω της αλλαγής ε, κυβέρνησης. Και Πρόσφατα παρουσιάσαμε πρόταση στο Συμβούλιο για, την, ε, για με την Αλβανία, την Βοσνία Ζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Ο οργανισμό επίση ε, σχεδιάζει να, ε, αποστείλει και στον Νίγηρα επιτετραμένου, πολύ σημαντική χώρα σε ό,τι αφορά την μεσογειακή οδό προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι η θέσπιση μια στρατηγικής διαδικασίας για την ε, ε, θέση σε ισχύ της ε, νέας ε, προσέγγισης που παρουσιάσαμε στις 29 Ιουνίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Θα θέλαμε όμως και εμείς να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να εμπλακεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο προπαρασκευαστικό στάδιο για να έχουμε ε, αυτή τη στρατηγική σε πραγματικό πολιτικό επίπεδο. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι η πραγματική ε, θέση σε λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, παραμένει μία από τι βασικέ προτεραιότητε τη Επιτροπή Γι' αυτό και κρατούμε αυτό τον μικρό κύκλο υποβολή εκθέσεων για να συνημερώνουμε συνεχώ, να πούμε πιέσει στα κράτη-μέλη. Θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση εκ του σύναγκης αυτής της κατάστασης, αλλά υπάρχουν πραγματικά πολύ θετικά πρώτα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Πρώτα τα μέλη πριν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω. Μπρίγκιτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα. Μιλήσατε για την έλλειψη στήριξης από πλευράς κρατών μελών. Μια στήριξη που έχει αποφασιστεί με τη νέα οδηγία περί της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Υπάρχουν λοιπόν ξεκάθαρα στοιχεία για το πότε θα φτάσουμε στο σημείο όπου και η τεχνική αρρωγή αλλά και τα ονόματα που αναφέρατε των 1500 συνοριοφυλάκων θα υπάρχουν όντως για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας ή είναι απλώς ε, κενές υποσχέσεις. Επίσης, μιλήσατε για την ε, υποστήριξη στον τομέα των επιστροφών. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα παραδείγματα για το τι ε, μορφή λαμβάνει αυτή η στήριξη. Είναι θέμα οργάνωσης, είναι πρακτική στήριξη για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Επίσης είπατε ότι ο αριθμός των επιστροφών αυξάνεται. Θεωρείτε ότι αυξάνεται γιατί στο παρελθόν τα κάτι μέλη δεν έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στις επιστροφές ή έχει αυξηθεί ε, η ετοιμότητα των χωρών προέλευσης να δεχθούν και πάλι πίσω τους υπηκόους ή υπάρχουν άλλοι παράγοντες που έχουν αυξήσει ε, τις επιστροφές. Κύριο Κάστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Έχω τις εξής δύο ερωτήσεις. Πρώτον, συνεργασία με τη Λιβική ακτοφυλακή. Τώρα συνεργάζομαστε και συνεργάζονται με το κράτος, αλλά υπάρχουν και εγκληματικές οργανώσεις ε, που δραστηριοποιούνται στον τομέα και, και συνεργάζονται με το κράτος επίσης. Ποια είναι λοιπόν η συνεργασία μας ε, με τις λιβικές αρχές και πόσο αξιόπιστε είναι τελικά αυτέ οι λογικέ αρχέ στη συνεργασία μα. Υπάρχουν παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τι συμβαίνει με τα πρόσωπα, τα άτομα τα οποία ε, συλλαμβάνονται καθοδόν. Ουσιαστικά θα ήθελα να δω τι συμβαίνει ε, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητε της ακτοφυλακής και αν υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, τοποθετεί αυτά τα άτομα στα σύνορα μεταξύ Λιβύης και Νίγηρα. Βέβαια, είναι κλειστά κάποια σημεία των συνόρων, όμως ε, πολλοί κόσμοι τα παρακάμπτει αυτά τα κλειστά σημεία. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι συμβαίνει και τι θα γίνει τελικά με αυτά τα σύνορα. Θα κλείσουν πραγματικά για να μην περνάει κανείς. Και τι δυνατότητες θα υπάρχουν να παρακάμψει κανείς αυτά τα ε, κλειστά σύνορα. Μάλλον παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Εδώ και ενάμεση χρόνο εγώ πήγα πριν από 1,5 χρόνο στα λιβικά σύνορα και είδα ε, την ε, βία της αστυνομίας. Δεν με ακούτε? Ναι, υπάρχει. Εντάξει. Μου λένε ότι υπάρχει ερμηνεία. Λοιπόν, ήμουν στα σύνορα στα βουλγαρικά σύνορα πιο συγκεκριμένα, πριν από 1,5 χρόνο. Και είδα την αστυνομική βία. I just thought I'd... I'd uh... Yeah, in, in French, my Swedish is perfect. But, okay, let's try. Από τα γαλλικά βγαίνει πολύ καλά η παρέμβασή μου. Τέλος πάντων, μιλήσω αγγλικά border uh, uh, in in Bulgaria, and I saw with my own eyes the uh, violence that that refugees had been subject to by border police. And I think that. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάσταση είναι η εξής. Εξακολουθούμε να έχουμε εκθέσεις. Διακόπτω την ομιλήτρια. Μα εγώ έχω... Α, τώρα δεν κλείνει το μικρόφωνο μου. Δεν κλείνει. Δεν κλείνει, δεν κλείνει.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 η ερώτησή μου είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και η Συνοροφυλακή για να ε, αυτέ αυτές τις περιπτώσεις και πώς, ε, ε, και πώς οργανώνονται οι κοινές επιχειρήσεις ε, μαζί με εθνικές ομάδες γιατί και για αυτές υπάρχουν εκθέσεις. Ποια, τι, σε τι έχουν οδηγήσει οι έρευνε σας. Θέλετε να απαντήσετε, ωραία. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις κυρία Ζίπελ. Για τα κράτη-μέλη. Ε, πιέζουμε να οριστούν και να ονοματιστούν ε, οι, ε, τα άτομα τα οποία θα ε, χρησιμοποιούνται εσείς το ζητήσατε παλιότερα στο τέλος των διαπραγματεύσεων για ποιο λόγο γιατί τότε που διαπραγματευόμασταν εσείς καταθήσατε σαφές ότι η πρόθεση του Κοινοβουλίου ήταν να διασφαλίσει ότι η ταχεία αντίδραση δεν θα ήταν απλώς μια υπόθεση εργασίας, αλλά θα αφορούσε άτομα τα οποία στην πράξη θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούν να κινητοποιηθούν σχεδόν αυτομάτως. Αυτό προσθέθηκε στις τελευταίες συναντήσει διαπραγματεύσεις για το, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Συνορφυλακής και Ακτοφυλακής. Πρέπει λοιπόν να περάσει το θέμα σε πολιτικό επίπεδο και τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη, ε, να ε, διορίσουν και να ονοματίσουν ε, αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό θα γίνει μέσω του Συμβουλίου, αν γίνεται, αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα τα οποία μας δίνει η συνθήκη. Όμω το θέμα δεν είναι αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι με τα ονόματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι ορίζονται θα έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς και θα διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προφίλ έτσι ώστε να καλύπτουμε όλες τι ειδικότητε και τις ανάγκες της ε, δύναμης ταχεία αντίδρασης. Αυτό θα το περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, το πολιτικό επίπεδο πλέον. Τώρα, για του ε, ε, για να δούμε τι συνέβη φέτος μέχρι τον Ιούνιο ας πούμε. Ε, η υπηρεσία έδωσε υποστήριξη σε 144 ε, επιστροφές, ε, επιχειρήσεις επιστροφών. Αυτό σημαίνει περίπου, ότι περίπου 7.000 άτομα τα οποία ήταν παρανόμως διαμένοντες 6.799 συγκεκριμένα επεστράφησαν στις χώρες τους. Αυτό δείχνει αύξηση 157% σε σχέση με πέρσι. Γιατί? Γιατί πρώτον ε, συνεχίζουμε και αυξάνουμε την πίεση που ασκούμε ιδιαίτερα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να δέχονται άτομα δικής τους προέλευσης οι οποίοι έχουν ε, εισέλθει παρανόμως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει απορριφθεί ε, η αιτησία ασύλου τους. 144 λοιπόν διαδικασίες επιστροφής έλαβαν χώρα προς τα Δυτικά Βαλκάνια, σχεδόν όλες, με τη δική μας υποστήριξη. Τι άλλο κάνει η υπηρεσία. Και αυτό δικαιολογεί και την αύξηση ορισμένων ε, ε, αύξηση επιστροφές και αποχώρηση μη Δυτικών Βαλκανίων. Αφορά τις δραστηριότητες πρώτης επιστροφής, δηλαδή διοργάνωση του ταξιδιού, ε, συνεργασία με τις ε, ε, χώρες επιστροφής για την ένταξη αυτών και με εταίρους σε τρίτες χώρες. Αυτό πρέπει να πούμε ενδεχομένω είναι ότι ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις επιστροφής μικρής μικρού διάστασης, μικρού μεγέθους γίνονται με εμπορικές πτήσει. Οι περισσότερε γίνονται με πτήσει charter. Αλλά αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούμε να διοργανώσουμε ένα πιλωτικό πειραματικό σχέδιο χρησιμοποίησης ε, εμπορικών ε, αεροπορικών εταιριών και θα πρέπει ιδιαίτερως να προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση για τρίτες χώρες μη Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Να διευκολύνουμε της διαδικασίας επιστροφής με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, στην ερώτηση Κιούστερ τώρα. Ε, την Τετάρτο πρωί νομίζω θα το συζητήσουμε. Γιατί ο ρόλος της υπηρεσίας ε, ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής ε, έχει σχέση με την ε, σε οκτωφυλακή της ε, Λιβύης η οποία έχει περιορισμένες αρμοδιότητες αλλά το συζητήσουμε την Τετάρτη νομίζω. Ε, πρέπει να πούμε τα εξή. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση που προσφέρουμε στην Λιβυακή εκτοφυλακή. έχουμε ένα μάθημα ένα σεμινάριο, ε, μάλλον στην εκπαίδευση αυτή υπάρχει και ένα σεμινάριο που διοργανώνει η Πατερμοστία του ΑΕΑ, για τους πρόσφυγες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεύτερον, τι θα πρέπει να γίνεται με αυτούς οι οποίοι μεταφέρονται στις λιβικές ακτές. Εδώ δίνουμε αρκετή χρηματοδότηση και στην υπατερμοστία και στον IOM για να λειτουργήσουν επί τόπου και να στηρίξουν την επανεγκατάσταση αυτών που χρειάζονται νομική προστασία ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα ζητήσαμε προσφορές από τα κράτη-μέλη και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν προσφορές για δυνατότητες επανεγκατάστασης από τη Λιβύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ε, τους πρώτους έξι μήνες αυτού του χρόνου ε, περισσότεροι έχουν επιστρέψει από τη Λιβύη στη χώρα προέλευσής τους ε, από ότι όλο το, προ, προηγούμενο έτος. Δηλαδή ε, προωθούμε τις εθελοντικές επιστροφές, ιδιαίτερα με χώρες, σε χώρες όπως το Μάλι και άλλες. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε μία συνολική προσέγγιση. Τώρα, για την Ιγυρία και τη Λιβύη. Ε, εδώ θέλουμε να ορίσουμε ένα ε, σύνδεσμο ε, με αυτές τις δύο χώρες από πλευράς μας. πολλά, έχουμε να, έχουν να γίνει στο Αγκαντές, από το οποίο ξεκινούν πολλές οδοί μετανάστευσης και εδώ εργαζόμαστε με την Πατιαρμιστή και τον IOM και θα συμπεριλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Νίγηρα ε, και χρειάζονται προστασία. Ε, επίσης, ε, εργαζόμαστε για την εθελοντική επιστροφή από το Αγκαντές στις διάφορες χώρες προέλευσης. Δύσκολα βέβαια μετράμε πολλές φορές το αποτέλεσμα. Έχουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι από 70.000 το μήνα έχουμε πέσει στις 12.500 μετανάστες από τον Ήγηρα. Επίση, προσπαθούμε να δώσουμε και κοινωνικο-οικονομική στήριξη ε, στην περιοχή του Αγκαντές ε, και στον Ήγερα γενικά προκειμένου να μειωθεί η ανάγκη να εργάζονται σε δίκτυα κινητών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς ε, άσκηση ε, στα βουλγαρικά σύνορα και εγώ ήμουν στη Σόφια πριν από δύο εβδομάδες ε, ήρθα σε επαφή με τον προσωπάρχη του ε, Πρωθυπουργού και με τον Υπουργό Δικαιοσύνη και ε, σχολίασα αυτό το θέμα με, μου ανέφεραν ότι έχουν λάβει μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθεί επανάληψη τέτοιου είδους ε, βίας και να τιμωρηθούν οι, οι υπεύθυνοι ε, θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, μερικές φορές, και θέλω να προσθέσω κάτι, ε, τα κράτη-μέλη, αν τα καταφέρουν και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε βάσει βάση την απόφασή μας για την φυλακή, πράγματι έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σημαντικό να μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε αποτελεσματικοί, κυρίως όσον αφορά αυτές τις ομάδες ταχείας δράσης. Αλλά πρόκειται και για ένα ε, κάπως γενικής φύσεως θέμα γιατί αποφασίζουμε εδώ, είμαστε με το Συμβούλιο, κάτι και μετά κράτη-μέλη αποφασίζουν κάτι διαφορετικό. Λένε, εντάξει υπάρχει ένας νόμος, αλλά εγώ ε, δεν θέλω να εφαρμόσω κάποια στοιχεία του νόμου. Αν το έκανα εγώ αυτός πολίτης, ε, ξέρετε πολύ καλά ότι θα υφιστάμει ταχύτατα τις επιπτώσεις. Εντάξει, δεν λέω να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πια έχω κουραστεί να υπάρχουν ε, οδηγίες που μερικές εξ αυτών είναι πολύ σημαντικές, δεν δείτε θέμα επ' αυτού, αλλά αν ε, δεν εφαρμόζεται τότε τι τις έχουμε. Γιατί γίνεται όλη αυτή η δουλειά. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να βρείτε λύση επ' αυτού, αλλά μια τελευταία συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί αναφερθήκατε, είπατε πολύ προσεκτικά, ότι κάποια κρατημέλη εφαρμόζουν τους κανόνες και το Συμβούλιο στο σύνολό του ε, θα έπρεπε ίσως να σκεφτεί κάποιες αντιδράσεις που προκύπτουν από τη συνθήκη. Ίσως να έχετε κατά νου ε, τη διαδικασία επί παραβάση που καλή είναι, αλλά σε τελική ανάλυση το να πληρώνει κανείς κάποια χρήματα αυτό δεν λύνει ε, το πρόβλημα. Εδώ δεν είναι το θέμα τα χρήματα. Βέβαια εντάξει δεν χρειάζεται να απαντήσετε γιατί και αυτό πολιτική δήλωση δική μου ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σύντομη θα είμαι. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, σχετικά με τις υποσχέσεις ε, περί επαναγκατάστασης που αναφέρατε, ποιος θα ε, κάνει τις αναφορές από τη Λιβύη, εσείς ή η πατερμοστία, γιατί στα δικά μου τα χαρτιά και δουλεύω αρκετά επ' αυτού, η η αρμοστία; δεν νομίζω ότι αναφέρει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Η Σόφη. Προκλήθηκα από αυτό που είπε η Μπίργκιτ και συμφωνώ απόλυτα μαζί της αλλά ίσως θα πρέπει και εμείς να αντιρωτηθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί για πολλά χρόνια απλά δεχτήκαμε να επισφραγίζουμε τις απόφυσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου και οποτεδήποτε υπάρχει δεν εφαρμόζεται. Ε, συστηματικά τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα και τα κράτη-μέλη αγνοούν το τι έχει αποφασιστεί, όχι μόνο για τη Λιβύη, αλλά σε πολλές επιτροπές. Και παρόλα αυτά όμως, ε, να ε, κάνουμε αυτό που μας λένε, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Τα κράτη-μέλη μετά λένε ότι ότι ή πολλοί λένε ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και αυτό γίνεται αδιάλειπτα και κάπως πρέπει να σταματήσει αυτό. Εάν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν θέλουν Ευρωπαϊκή Συνεργασία, να μας το πούν. Να σταματήσουμε να ε, παίζουμε με το δικό τους το βιολί. Άλλος παρακαλώ πριν δώσουμε το λόγο στον Σάιμον. Όσον αφορά το θέμα της επαναγκατάστασης, κοιτάξτε δεν είμαι και ο πιο καλός εμπειρογνώμων, αλλά νομίζω η πατιαρμοστία θα προτείνει τα ονόματα. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την επαναγκατάσταση. Ήμουνα πρόσφατα στη Γενέβη, συζήτησα με τον Πολκετόρκ και νομίζω ότι η προετοιμασία γίνεται σε συνεργασία με την Τερμοστία. Το θέμα είναι κατά πόσον η Τερμοστία είναι σήμερα σε θέση να τα κάνει όλα αυτά, γιατί η κατάσταση της ασφάλειας είναι διαφορετική, αλλά το θέμα και η πρόθεση είναι να συνεργαστούμε μαζί τους. Για τα επόμενα θέματα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, να πω μόνο ότι γνωρίζουμε πολύ καλά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα ε, των συνθήκων και του τελευταίου μήνε έχουμε δείξει ότι θέλουμε να λάβουμε και να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα οποτεδήποτε ε, προκύπτει ε, παραβίαση των συνθήκων, Ουγγαρία, η αποτυχία των κρατών μελών να εφαρμόσουν νομικά δεσμευτικές αποφάσεις μετεγκατάστασης. Δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε ο διορισμός εμπειρογνωμόνων. Νομίζω ορισμένα κράτη-μέλη σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων δεν έχουν καταλάβει αυτό που είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις. Ότι δηλαδή εδώ δεν διακυβεύεται η, η υποθετική αναφορά ονομάτων, αλλά διακυβεύεται περισσότερο το να υπάρχει ένα πουλ ταχείας αντίδρασης, ένα φετρικό, μια τέτοια φετρική δύναμη. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η επόμενη φάση είναι να στείλουμε ένα μήνυμα σε πολιτικό επίπεδο στους υπουργούς υπενθυμίζοντας την πρόθεση του Κοινοβουλίου ε, όταν εγκρίθηκε η σχετική νομοθεσία και μετά ελπίζω να προκύψει αυτή η τομή που όλοι επιθυμούμε διακόσμια. Πάμε τώρα ε, στο επόμενο σκέλος της συζήτησης που αφορά στη Συμφωνία για την Αποστολή Ομάδων Σύνορο Φυλακής στη Σερβία. Και αυτό πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ίσως μπορούν να μείνουν οι βουλευτές, ε, και οι νομικοί σύμβουλοι, οι συγητές, εκπρόσωποι του Προεδρείου, νομική υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος δεν είναι αρμόδιος, παρακαλώ να φύγει από την αίθουσα. Αν δεν είσαι σε τον κατάλογο που διάβασα, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να φύγετε. Ευχαριστώ.